Γεια σας, συνάδελφοι. Ξαναρχίζουν οι εργασίες της Επιτροπής μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον Γενικό Γραμματέα Αλίας της Ισπανικής Κυβέρνησης. Με αγάπη του απευθύνουμε χαιρετισμό τον ευχαριστούμε που ήρθε στις εργασίες μας. Και αμέσω περνώ σημείο 9. Ανταλλαγή απόψεων με τον ε, κύριο Καρέλ Ντεγκούχτ, Ευρωπαίο Επίτροπο φθηνό για θέματα εμπορία. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε που είστε εδώ. Από το βάθο τη καριάς μου. Διότι από τη στιγμή που όπως ξέρετε όλοι προγραμματίσαμε την ε, παρουσία του στην Επιτροπή, μας το είπε αμέσως και μας επιβεβαίωσε ότι θα έρθει. Πράγμα το οποίο δεν κάνουν και κάποιοι άλλοι επίτροποι που είναι ίσως και πιο κοντά στα θέματα της Επιτροπής μας. Εξ ονόματος λοιπόν της Επιτροπής μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Για ποιο λόγο θέλαμε να είστε εδώ, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είδα τον Επίτροπο και του είπα τι ακριβώς ενδιαφέρει την Επιτροπή μας. Το επαναλαμβάνω όμως σύντομα. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να ξέρουμε είναι οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ε, υπογράφονται ή θα υπογραφούν όπως ξέρετε πολλά από αυτά έχουν μεγάλη σχέση με τον Αλία και με την ε, μεταποίηση των προϊόντων της αλίας σε όλη την Ευρώπη. Μιλώ για τις παρούσες συμφωνίες και για τις μελλοντικές. Και θα θέλουμε πάντα να έχουμε με τη γενικότερα, με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, μία πάρα πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων να επικοινωνούμε ώστε να ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο, να μην έχουμε αποκλήσεις απόψεων αν μπορούμε να το επιτύχουμε. Γι' αυτό θέλουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ Μπορείου και της Γενικής του Διεύθυνσης της ίδιας της Επιτροπής Εμπορίου ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και ημών να υπάρχει πάρα πολύ καλή και εύρυμη σχέση. Έχουμε να σας κάνουμε πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Μας ενδιαφέρουν οι διάφορες συμφωνίες που υπάρχουν με χώρες της περιοχής ΑΣΕΑΝ, με το Βιετνάμ, με την Ιαπωνία. Γι' αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε. Σας δίνω το λόγο κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ και πάλι που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. για την πρόσκληση στη σημερινή σας ε, συνεδρίαση. Το διεθνές εμπόριο έχει ιδιαίτερη σημασία από διάφορες πλευρές για την Αλία. Αντίστροφα, η Αλία έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε διμερές και πολυμερές επίπεδο ε, κατά τη διάρκεια διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων ε, και θα μας απασχολεί αυτό η συζήτησή μας και πιστεύω ότι αμφότεροι θα είμαστε ειλικρινείς. Θεσμικός πώς αρμόδια είναι η κυρία Δαμανάκη, αλλά η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ και η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου συνεργάζονται σε καθημερινή βάση πολύ στενά για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μόλις γευμάτισα με την <laughs> κυρία Δαμανάκη φάγαμε ψάρι, πρόεδρε. Το θέμα είναι που είχε ψαρευτεί το ψάρι που φάγαμε. Και τι είδος ήτανε. Πιστεύω ότι μάλλον καλό ήταν. Έτσι νομίζει η Επιτροπή, ακούστηκε ένα σχόλιο εκτός μικροφώνου. Καλό είναι όμως που σκέφτεται η Επιτροπή, απαντάει ο Επίτροπο, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι δεν συνέβαινε πια αυτό. Λοιπόν, ε, για τα εμπορικά ζητήματα και συγκεκριμένα στον τομέα Λίας, ποια είναι τα ζητήματά μας. Ε, ο γύρος ε, των διαπραγματεύσεων της Ντόχα έχει σταματήσει εδώ και καιρό, όπως γνωρίζετε, με λίγες προοπτικές να συνεχίσει στο προσεχές μέλλον, εκτός για τα μέτρα διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε επισταμένα σε συνεργασία ε, με διάφορες χώρες που ακολουθούν το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης για τη διαχείριση των στόλων μας και για τις πολιτικές ανάκτησης αποθεμάτων. Ε, ε, ε, μία συμφωνία συνυπογράφηκε το 2010 με την Κορέα, με τη Σιγκαπούρη θα υπογράψουμε τη συμφωνία μέχρι το τέλος του 2012, ακολουθεί και η συμφωνία με την Μαλαισία και αρχίσαμε διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ και ενδεχομένως το 2013 με την Ταϊλάνδη. Ελπίζουμε δεν να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και η Ινδία είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό εταίρος στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως είναι χρονοβόρες οι διαπραγματεύσεις. Ε, και υπερβαίνουν συχνά τη θητεία ενός Επιτρόπου Αρμοδίου για τα θέματα εμπορίου. Τώρα πηγαίνω στην άλλη Ήπειρο, την Αμερική, συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, έχουμε προκεχωρημένες διερευνητικές πρωτοβουλίες για τη σύναψη διμερού συμφωνίας με τη ΣΥΠΟ. Ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Κολομβία, το Περού και την Κεντρική Αμερική. και στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο το Δεκέμβρη αναμένεται η επικύρωσή τους από το Κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε δε και τις συζητήσεις με τον Μερκοσούρ Ισμάτιν προς το παρόν. Ε, Είμαστε απασχολημένοι με την Γεωργία, την Μολδαβία και την Αρμενία και με τις μεσογειακές χώρες. Ε, οι διαπραγματεύσεις για τις ε, οικονομικού χαρακτήρα συμφωνίες μας απασχολούν και μας απορροφούν πολύ χρόνο. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα έχουμε αποκομίσει τα ωφέλη από τις ενδιάμεσες οικονομικές συμφωνίες των χωρών που δεν έχουν υπογράψει ή επικυρώσει αυτές τις συμφωνίες. Έχει παρέλθει μία πενταετία και γνωρίζω τις ανησυχίες σας κυρίως για τη συμφωνία με την Παππούα Νέα Γουινέα. Θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Δεν έχουμε ουδόλωσε την ε, πρόθεση να συμπεριλάβουμε τον κανόνα ε, της ε, προέλευσης πέρα από τον ειρηνικό θα αποκομίσουμε εδώ και κάποια ωφέλεια από την παγκόσμια ανάπτυξη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Θα πρέπει να δράξουμε αυτές τις ευκαιρίες ε, γιατί διερχόμαστε μια κρίση άνευ προηγουμένου και έχουμε πλήρη επίγνωση του ότι κάποιες ε, συμφωνίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τα θέματα αλίας. Ε, Καναδάς με μονομένα μέλη του ΑΣΕΑΝ, χώρες ΑΚΕ και Λατινική Αμερική. Το θέμα των επιθετικών και των αμυντικών συμφερόντων μας μας απασχολεί διαρκώς και επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την αλία. Χρειαζόμαστε εισαγωγές ε, προϊόντων ε, για να καλύψουμε τα δύο τρίτα της κατανάλωσής μας, οπότε οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, οι περίφημες FTAs, μπορούν να τονώσουν την ανάκαμψη, να φέρουν νέες επενδύσεις στον κλάδο της αλίας για να επιτύχουμε τους στόχους περιβιωσιμότητα. Τα αλλιευτικά προϊόντα ε, συνιστούν ένα περατό πόρο και πρέπει να κάνουμε προσεκτικές επιλογές με τρόπο ώστε να καλύψουμε τις όσες ανησυχίες και προβλήματα υπάρχουν σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, Έχουμε κατά νου ότι η αντιαγωνιστικότητά μας για κάποια προϊόντα, παραδείγματο χάρη τόνος, σε κονσέρβα, ε, ε, εξαρτώνται από τους δασμούς ε, και κυρίως από την οικονομική ανάπτυξη κάποιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υστερούν. Θέλουμε να προστατεύσουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων τα συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως Επίτροπος Εμπορίου ε, δεν θεωρώ ότι είναι δόγμα και αυτός σκοπός το να τονώνουμε το διεθνές εμπόριο αλλά χρησιμεύει στην τόνωση της αλλιευτικής βιομηχανίας βρίσκοντας μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. δεν επικύρωσε το Κοινοβούλιο τη Συμφωνία με την Παπουασία Νέα Γουινέα αλλά αυτό που έγινε είναι ότι δημιούργησε δημιουργήθηκαν χάρη σε αυτή την συμφωνία νέες θέσεις απασχόλης και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις σωστές επενδύσεις τα, οι πρώτες ύλε, δηλαδή προϊόντα φινοειδών, μπορούν να εξαχθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προτού ε, μεταποληθούν ως επεξεργασμένα προϊόντα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπραγματευόμαστε με τον Καναδά για την άρση των εξαγωγικών περιορισμών για αλλιευτικά προϊόντα για κάποιες από τις περιφέρειες και τις Κομιτείας ε, του Καναδά. Επίση ε, θέλουμε πρόσβαση στου καναδικού ε, λιμένε για τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα θέματα σχετίζονται με συμφέροντα των οικονομικών φορέων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ενίσχυση τη διεθνού παρουσία του. Οι κρατέ τέτοιε συμφωνίε προσελκύουν επενδύσει και προστατεύουν καλύτερα τι επενδύσει. Επιστεύω ότι δεν προβάλλεται αρκετά αυτή η διάσταση, γι' αυτό και την αναφέρω εγώ σήμερα σήμερα. Ε, χρησιμοποιούμε τις συμφωνίες συγκεκριμένα ως πλατφόρμες, ώστε οι εταίροι μας να συνεργαστούν μαζί μας για θέματα βιωσιμότητα και τα συμφέροντα. Δεν θέλουμε ε, να τα περιορίζουμε στις οικονομικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Παρακινούμε του εταίρου μα να συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα και να καταπολεμούν την παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία. Χρησιμοποιούμε τι διαπραγματεύσει, είπαμε, χρησιμοποιώντα ω πλατφόρμα τον ειρηνικό για να ε, επιτύχουμε βιώσιμη αλία, βιώσιμη διαχείριση τη αλία και αυξημένη διαφάνεια. Τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, ε, κάποιες εμπορικές διαπραγματεύσεις ε, μας προσφέρουν μια πλατφόρμα βήμα συζητήσεων για, για την πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους, ε, παραδοσιακός πως δεν μπίπτουν στη ναι, διαπραγματευτική μας εντολή αυτά τα θέματα, αλλά αυτό άλλαξε πρόσφατα και το κρίνουμε κατά περίπτωση Πίνε στην περιοχή του Ειρηνικού Ακολουθήσαμε αυτή τη γραμμή διότι θεωρήσαμε ότι οι εταίροι μας ήταν επίσης έτοιμοι να διαπραγματευτούν για αυτά τα ζητήματα. Είμαστε σε αρχικό στάδιο βεβαίως, αλλά είναι πολλά υποσχόμενες οι διαπραγματεύσεις και με συγκεκριμένα ε, θα, οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε οικονομικές συμφωνίες. Δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίζουμε τη σημασία των διεθνών εμπορικών μέσων. Καλωσορίζεται το, τη μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων GSP ε, προσφέροντας περισσότερο ωφέλη στις χώρες που τα χρειάζονται περισσότερα. Είναι πάρα πολύ νωρί ε, για να δούμε ε, ποιο, ποια χώρα είναι επιλέξιμη για τις επιδοτήσεις το, για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων αλλά εξαγωγικές χώρες είναι επιλέξιμες και Αυτές θα προτιμήσουμε για την διαπραγμάτευση ε, ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, ούτως ώστε να προωθήσουμε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να είναι επωφελές και για τους δικούς μας οικονομικούς φορείς. Χρησιμοποιούμε μέσα διεθνούς εμπορίου επίσης για να τονώσουμε την βιώσιμη ελεία. Μιλάω για την, το μέσο καταπολέμησης της ε, παράνομης ε, λαθρέας και αναρχής ε, αλίας που επιτρέπει την επιβολή σοβαρών κυρώσεων. Αναφέρομαι στο εργαλείο, στο μέσο που πρόσφατα σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε για τη διαχείριση των κοινών αλλιευτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρε, όπως είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου, χάρη στη σημερινή συζήτηση μπορούμε να τονίσουμε τους ε, δεσμούς ανάμεσα στην ε, πολιτική αλλίας και την πολιτική διεθνούς εμπορίου. Νομίζω ότι ξεκαθάρισα πως ε, δεν υπάρχει μία μονοδιάσταση στο θέμα. Παντού υπάρχουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις και αντιμέτωπος με όλα αυτά και με την ιδιότητα του Επιτρόπου Αρμοδίου για τα εμπορικά ζητήματα προσπαθώ να εξισορροπήσω πάντοτε τις απαιτήσεις με τα συμφέροντα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ταυτόχρονα θεμητές προσδοκίες του ε, κλάδου της αλίας και επιταγές της πολιτικής αλίας που πρέπει να σεβαστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα κάνουμε τώρα ένα πρώτο γύρο παρεμβάσεων. Θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στους συντονιστές και μετά στους άλλους συναδέλφους. Αρχίζουμε με το ΕΛΚ. Δεν είναι εδώ συντονιστής, αλλά δίδω το λόγο στην κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο Ντεγκούχ. Χαίρομαι και σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα για να μας εξηγήσετε και να κάνετε σχόλια και παρατηρήσεις για τα θέματα που μας απασχολούν, κυρίως την αλληλεία σχέση με το εμπόριο. Μας είπατε, θα κάνω ένα σχόλιο και μετά συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μας είπατε ότι η Ελία είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της Εμπορικής Επιτροπή Πολιτικής. Όντως, εγώ νομίζω ότι θα επικεντρωθώ σε αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό στον τομέα της Αλίας. Δηλαδή, η εμπορία των θηνοειδών και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όπως ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε για αυτό το είδος 42 εκατομμύρια τόνους. Η παραγωγή κονσέρβας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 7% της παγκόσμιας παραγωγής κονσέρβας και η κοινοτική ε, λοιπόν ε, Κοσερβοποίηση στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ μικρή και πολύ λίγα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Οτιδήποτε όμω κάνουμε στο εξωτερικό μπορεί να επηρεάσει άλλε χώρε με τις οποίες στο παρελθόν είχαμε πάρει κάποια μέτρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο και εμάς μας ανησυχεί. Μην πιστεύετε ότι εμεί εδώ απλώ και μόνο είμαστε εδώ υπερασπίσουμε αυτή την ελάχιστη παραγωγή, τι στρατηγικές μπορούμε να υιοθετήσουμε χωρίς να γίνουν πάρα πολύ ακραίες ε, κινήσεις όπως είχαν γίνει τις άλλες τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το θέμα της παπαζίας Νέας Γουινέας. Ξέρουμε ότι ε, επηρέασε τις Αιχέλες. Θα Ξέρουμε ότι τότε υπήρχε επιρροή της πολιτικής με τη μια χώρα την άλλη. Τι θα γίνει τώρα με την Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη είναι η πιο ανταγωνιστική χώρα όσον αφορά την κονσερβοποιία θηνοειδών. Εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, αλλά ό,τι γίνει με την Ταϊλάνδη θα επηρεάσει την Παπουαζία Νέα Γουινέα. Την Παππούα με συγχωρείτε Νέα Γουινέα. Τώρα, όταν έχουμε μηδενικούς δασμούς, στην περίπτωση της Αυστραλίας και άλλων χωρών, της Ταϊλάνδης και άλλων χωρών, η Παπό είδε ότι δεν είναι ανταγωνιστική. Και έτσι έστρεψε τις ε, εξαγωγές της προς εμάς, για να είναι πιο ανταγωνιστική. Αυτό με απασχολεί. Όλες αυτές οι απότομες αλλαγές να ληφθούν υπόψη. Διότι αυτό το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις για την Παπούα μπορεί να επηρεάσει τις Ειχέλες και αυτό που κάνουμε με την Ταϊλάνδη και την ε, Βιετνάμ και πάλι μπορεί την Παπούα να την ε, ε, επηρεάσει. Τώρα, με τα θέματα του ειρηνικού. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεστε τα θέματα ΕΠΑ με άλλες χώρους που είναι στην Forum Fishery Agency που ζητούν ε, περισσότερα λιευτικά σκάφη. Θα ήθελα λοιπόν, και εγώ μίλησα με τη Γενική Διεύθυνση Μάρε, να σας ζητήσω το εξής. Θα μπορούσε να υπάρχει ε, εστίαση στα περιφερειακά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Είχατε πει στην ε, Επιτροπή Trade όταν συζητούσαμε για την Αγουινέ ότι είχαν ε, δοθεί κάποιες δυνατότητες αλίευσης οι οποίες εκ των υστέρων απερίφθησαν. Όταν ε, λοιπόν ασχολούμεθα με διαπραγματεύσεις που αφορούν όλες τις χώρες του Ατλαντικού, του Ειρηνικού, μπορείτε να κάνετε εκ παραλίλου διαπραγμάτευση λαμβάνοντας υπόψη τι έχει γίνει και σε περιφερειακό επίπεδο από άλλους, όπως έκαναν οι ΙΠΑ Φερρυπίν, συγκεκριμένη περίπτωση, για να μπορούν να αλλιεύουν στις περιοχές αυτές. Επίσης, αυτό θα ήθελα να σας πω, για θέματα αλληγίας, αλλιές, κάνετε ε, άστε λίγο στο περιφερειακή κατάσταση και προβλήματα που υπάρχουν. Και η ερώτησή μου, πιο συγκεκριμένη, είναι τι σκέφτεστε για αυτό που σας λέω, να εστιαστείτε δηλαδή σε περιφερειακές ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Ποια είναι η γνώμη σας. Ποια είναι η πρόοδος που βλέπετε στην ε, ΕΠΑ του Ειρηνικού. Με ποια ταχύτητα προχωρούν τα πράγματα. Και μπορείτε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει με την Ταϊλάνδη, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι η πιο ανταγωνιστική χώρα σε θέματα κονσερβοποίησης θηνοειδών. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται μπορούν να επηρεάσουν άλλες χώρες. ΑΣΕΑΝ, ΑΚΕ και με ανησυχούν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θα ήθελα η στρατηγική που ακολουθείτε να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στις ε, ε, χώρες της περιοχής, κυρίως με την ε, του τόνου. Ποια ήταν ε, η τελευταία ερώτηση? η Συμφωνία ελευθέρω μπορεί με την Ταϊλάνδη. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε αυτή τη στιγμή να μου πείτε κάτι περισσότερο. Να μου πείτε δηλαδή πώς ε, διεξάγεται ο διάλογος. Εμένα με αφορά μόνο τι συμβαίνει με την ε, Αλία. Οι άλλοι τομεί δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά για την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ θα ήθελα να έχω κάποιες πληροφορίες. Και μετά τι γίνεται με το ΕΠΑ στον Ειρηνικό. Υπάρχουν δυνατότητες διεύρυνσης της συμφωνίας και σε με ποιο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή η δική σας οπτική γωνία και αυτή της Μάρε ποια είναι για αυτά τα θέματα τα οποία σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρόντους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πολλές ερωτήσεις για να σας πω την αλήθεια η κυρία Φράγκα ουσιαστικά ανέφερε τις πιο σημαντικές όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ. Φυσικά αυτό που θέλουμε είναι να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Από την άλλη έχουμε υψηλά πρότυπα, ε, θέλουμε να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύεται το περιβάλλον στον τρόπο αλληλείας και όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εμπορικές μας συμφωνίες πολλές φορές ε, ερχόμαστε σε αντίθεση και εδώ εντό τη Επιτροπής για επιμέρου συμφωνίε. Όπω είπα, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τι απαιτήσει μα Τώρα, εσείς πού διαβλέπετε τις περισσότερε δυσκολίε όσον αφορά τα επίπεδα που διαβλεπετε τι περισσοτερε δυσκολιε οσον αφορα τα επιπεδα που προβλεπουμε και ε, αυτό έχει αποτελέσει ζήτημα και για την Επιτροπή Γεωργίας και θα ήθελα να μου πείτε πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση, να φροντίσουμε να μην απολέσουμε ανταγωνιστικότητα αλλά ταυτόχρονα να τηρούμε τα επίπεδά μας. Πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Ε, έχουν υπάρξει πολύ ζωντανέ συζητήσει, τόσο εντό Επιτροπή όσο και εντό τη δική μου πολιτική ομάδα. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε μια απάντηση γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριο Γκάλεχερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Επίτροπο και να τον ευχαριστήσω για τις απόψεις μας παρουσίασε ως ε, Επίτροπος Εμπορίου. Και φυσικά υπάρχει ένας ανάποσπαστος δεσμός μεταξύ του εμπορίου και της ελίας. Και φυσικά γνωρίζουμε όλοι, κοιτώντα τα στατιστικά στοιχεία του εμπορίου για τι εισαγωγέ και τι εξαγωγέ, ότι εισάγουμε λόγω ανάγκη φυσικά υπερβολικά πολλά ψάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και φυσικά ο μόνο τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε θα είναι να βεβαιωθούμε ότι η κυρία Δαμανάκη θα μεριμνήσει ώστε να έχουμε ε, βιώσιμη αλληλεία αλλά επιπλέον και έλεγχο των καλλιεργιών. Πράγματι, οι εισαγωγές διατηρούν ένα στατουσκό και έχουμε μια ευθύνη να φροντίσουμε να γίνουν όλες οι προσπάθειες υποστηριξής τους. Πάντα όλοι κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ουσιαστικά εγώ θεωρώ υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για τις καθυστερήσεις και για τη διεκπαίρεωση των αιτήσεων για ε, ηχθειοκαλλιέργειες. Θα έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία μία στάση. Υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εμπορικές, ε, αληφτικές. Κύριε Επίτροπε, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό που θα σας πω τώρα και κατά πόσο είστε αρμόδιος γι' αυτό μπορείτε να μας το ενημερώσετε. Εγώ επισκέφθηκα τη Γρυλανδία πρόσφατα και μίλησα ε, εκεί με τον πρόεδρο για τις αντιπροσωπές για τις αρκτικές χώρες και μου είπαν ότι μιλάμε για χιλιάδες ε, γνωρίζουν όλοι ότι τα λευκά προϊόντα αποτελούν μεγάλο ε, ε, μεγάλο πόρο για τις χώρες αυτές ε, και για τους ε, ηθαγενείς, για τους αυτοχθόνες, συγγνώμη. Και υπάρχει μια προσφυγή των Καναδών στον οργανισμό εμπορίου και για τα δέρματα φώκιας και ξέρουμε πότε αναμένουμε μια απάντηση. Επίσης αναφέρατε εμπορικές κυρώσεις. Δεν ξέρω τι άποψη σε σχέση με τις κυρώσεις, διότι εμείς είμαστε υπέρ μιας ελεύθερης οικονομίας, αλλά έχουμε ε, κάποια σημαντικά προβλήματα. Όπως μη αηφόρο αλληλεία σε πόρους και σε δικά μας υδάτα, αλλά και σε αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα. Δεν θέλω να αναφέρω μια συγκεκριμένα χώρα, γιατί όταν μας έκανε η Επιτροπή την πρόταση να επιβάλλουμε κυρώσεις, εμείς θεωρούσαμε ότι δεν ήταν αρκετά ισχυρές είδαμε σε κάποια παραδείγματα ότι 90-95% των συγκεκριμένων ηχθείων ε, εξάγονταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς δεν σήμαινε και τίποτα ιδιαίτερο. Θέλω να μου πείτε δηλαδή τι γίνεται με τις εμπορικές κυρώσεις. Πώς πιστεύετε εσείς ε, ως Επίτροπος ε, Εμπορίου. Είμαι σίγουρος ότι πώς ε, έχουν οριστεί αυτέ οι εξαιρετικέ περιστάσεις. Είμαι σίγουρο ότι συμμετείχαν. Κάποια τέτοια μέτρα μπορεί να επηρεάζουν το εμπόριο ή κάποιες άλλες πτυχέ του εμπορίου. Θα πρέπει να μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα πάρουμε ή όχι μια απόφαση. Ελπίζω λοιπόν τα εργαλεία που εμείς έχουμε δώσει στην Κομισιόν ομόφωνα, νομίζω μόνο εννέα βουλευτές ψήφισαν κατά. Θα θέλαμε λοιπόν την άποψη του Κοινοβουλίου να αντικατοπτρίζεται στι εργασίε τη Κομισιόν. Θα θέλαμε να το λάβει υπόψη του κύριο Επίτροπο και να ε, γνωρίζει ότι υποστηρίζουμε πλήρω τον Επιτροπό Εμπορίου και του υπόλοιπου. Η κυρία Λέβεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ ω συντονίστρια των Πρασίνων. Σα καλωσορίζω εδώ και ειδικά επειδή είμαι εισηγήτρια της έκθεσης ε, για τη μεταρρύθμιση της ε, εξωτερικής κοινή ελληνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Όντας λοιπόν η συγγήτρια αυτής της έκθεσης ε, πάντα διαβλέπω τον κίνδυνο ότι προσπαθούμε η στόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι βιώσιμη στο μέγιστο βαθμό δυνατό η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί συμφωνίες μόνο με χώρες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν κρατούς δικαίου, εργατικά δικαιώματα, που πληρούν όλα τα πρότυπα τα οποία απαιτούμε και εμείς από το δικό μας στόλο, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ε, αναμένουμε να πληρούν οι στόλοι μας. Ενώ ταυτόχρονα, όπως είπατε κύριε Επίτροπε, εισάγουμε τα δύο τρίτα της όλης κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάθε ψάρι που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, αλλιεύεται ε, βιώσιμα, διότι διαφορετικά απλά μετακυλούμε τα προβλήματά μας σε κάποιον άλλο. Τα προβλήματα εκμετάλλευσης, το, υπερβολικής εκμετάλλευσης των αποθεμάτων, υπεραλίευσης, ε, ε, υποβάθμισης των κοινωνικών ε, επιπέδων. Τα ψάρια δεν είναι αγαθό, είναι αγρία ζώα, είναι κομμάτι της φύσης, αλλά είναι και τροφή. Πάντα μιλάμε λοιπόν και για τη διατροφική ασφάλεια πολλές φορές εδώ, σε, την ασφάλεια των τροφίμων σε διάφορες χώρες όταν ε, συνάπτουμε συμφωνίες αλληλευτικές με ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όλοι οι επίτροποι ανάπτυξης, εμπορίου και αλίας θα πρέπει να συνεργαστούν με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος για αυτά τα ζητήματα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε μια παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για μια νέα λίστα χωρών κατ' εξαίρεση που δεν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού κατά της παρανομής λαθρέας και ανεξελίας. Οκτώ τέτοιες χώρες έχουν αναγνωριστεί και έξι, μετά από έξι μήνες θα έχουμε πιθανώς εμπορικές κυρώσεις κατά αυτών των χωρών. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς κύριε Επίτροπε είναι τι άποψη έχετε εσείς για αυτή τη λίστα και πώς συνεργάζεστε με την Επίτροπο κύριε Δαμανάκη σχετικά με αυτή τη λίστα. Επίσης αναρωτιέμαι πως για παράδειγμα στην εμπορική συμφωνία με την Κορέα όπου αναφέρατε και το αληφτικό της κομμάτι. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε εισαγωγές από την Κορέα παρότι γνωρίζουμε ότι η Κορέα είναι γνωστός τόπος παράνομης λαθρέας και αναρχής αλίας. Ε, διάφορες ε, περιπτώσεις γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή με εκκρεμόντα πρόστιμα που δεν έχουν πληρώσει εταιρείες, οι κορεατικές εταιρείες θα με ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσω την άποψή σας επί του θέματος και για πιθανές εμπορικές κυρώσεις κατά της Κορέας. Εάν η Γενική Διεύθυνση Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έχουν, έχει συζητήσει με τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για την Κορέα ως μη συνεργαζόμενη χώρα, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω λάβει εγώ από κάθε πηγή, η Κορέα δεν είναι συνεργάσιμη, δεν έχει καν σύστημα VMS πάνω στα σκάφη της Συνεπώς δεν μπορούν να δώσουν καμία διασφάλιση για τις ε, δραστηριότητες των στόλων μεγάλων αποστάσεων και Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Και τέλος, κυρία Φράγα, ανέφερε εμείς στην Παπονία Γουινέα τη σχετική συμφωνία και εσείς ε, ε, αναφέρατε την ΕΠΑ με την Παπονία Γουινέα ναι, και την εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης, στο, καταγωγή στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που θα ήθελα να σας συστήσω. Ονομάζεται Can Paradise και δείχνει τις επιπτώσεις που είχε αυτή η συμφωνία στον τομέα της και στον τοπικό πληθυσμό στην Παπανέγου Νέα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πραγματικά δεν έχει ωφελήσει ιδιαίτερα τους ε, τοπικούς αλληλείς ή τον τοπικό πληθυσμό στην Παπανέγου Νέα Αντιθέτως υπήρξαν πολλές ε, καταχρήσεις γης ε, από ξένες εταιρείε ε, για δραστηριότητες παραγωγής διαφόρων προϊόντων βασισμένων στην αλληλεία, επίσης πορνεία, εκμετάλλευση εργαζομένων. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Λέβεν. Κύριος Φερέρα. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίαση που έκανε. Σίγουρα θα είχατε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις προτάσεις Επιτροπής Αλίας ή γενικότερα του Κοινοβουλίου για ζητήματα που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο και την αλία. Και σίγουρα θα γνωρίζετε και την πολύ σημαντική έκθεση που ανέκρινε το Κοινοβούλιο, την έκθεση του συναδέλφου Καντέκ από το ΕΛΚ, το οποίο το κεντρικό μήνυμα ήταν το εξής. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τον ευρωπαϊκό αλλιευτικό κλάδο στο βωμό του ελευθέρου εμπορίου. Ε, είναι πάγια θα έλεγα θέση της Επιτροπής μας και εγκαρσίως πως ε, παρατηρείται και σε άλλα σε άλλες πολιτικές ομάδες ε, και στις παρεμβάσεις των προλαλισσάντων διεφάνει ξεκάθαρα η ανησυχία αυτή. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στην Ευρώπη, στην Αλία. Είναι το πρόβλημα των αμοιβών το θέμα των τιμών. Ε, ε, υπάρχει μεγάλη πίεση στην, πρώτη, στην τιμή της πρώτης μεταπόλησης που είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Οι τιμές αυτές ε, απειλούν κυρίως τα τμήματα του στόλου μικρής κλίμακας, εραστεχνική αλληλεία, παράκτια αλληλεία και όπως γνωρίζετε εκπροσωπούν αυτοί οι δύο κλάδοι μεγάλο τμήμα του κλάδου της αλίας. Πιέζονται προς τα κάτω λοιπόν οι τιμές της πρώτης μεταπόλησης και ταυτόχρονα διαβρώνονται σε μεγάλο βαθμό τα εισοδήματα των επαγγελματιών του κλάδου. Όπως ακούσαμε από τους συναδέλφους, Ε, γίνονται εισαγωγές αλλιευμάτων από χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους δικούς μας κανόνες ε, στον τομέα του περιβάλλοντος, ε, ως προς το, εργατικό δίκαιο κτλ. κτλ. Όταν λέμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε την αλληλεία στο βωμό του ελευθέρου εμπορίου, αυτό εννοούμε που μόλις σας περιέγραψα. Επίτροπε, εσείς συχνά μα κάνετε, ε, μας απαγγέλλετε μανιφέστα, αν θέλετε, του ελευθέρου εμπορίου και οφείλετε να διαπιστώσετε όμως τις αρνητικές επιπτώσεις απελευθέρωσης του εμπορίου, κυρίως στον τομέα της αλίας ε, Και σε κάποιες από τις εμπορικές ε, συμφωνίε που τώρα διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερο βάρος η αλία με την Καναδά, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, με τις ασιατικές ε, χώρες και τις χώρες ΑΚΕ συγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Σε κάθε μία από αυτή τη συμφωνία που προαναφέρατε και στο ε, αλληλευτικό τμήμα τους, ποια προβλήματα διαπιστώσατε και ποιες ε, διαφορές με τους εταίρους μας διαπιστώσατε πάλι για το κομμάτι της αλίας. Μιλήσατε για τα αμυντικά συμφέροντά μας. Έχουν αναφερθεί ρητά σε κάθε μία από αυτές τις συμφωνίες ε, που διαπραγματεύεστε. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Α, και για τις χώρες ΑΚΕ. Και ε, μία τελευταία ερώτηση. Γνωρίζουμε το τέλμα στο οποίο έχουμε περιέλθει λόγω της αυξημένης αντίστασης που δείχνουν πολλές από αυτές τις χώρες για την ε, ε, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα σύντομο απολογισμό ε, των συμφωνιών που ε, δεν μπορούν πλέον να προχωρήσουν, κυρίως σε σχέση με την Αλία. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ σύντομα. Μου ζήτησε και ο κύριος Τόρβαρ την συζήτηση μετά τους συντονιστές. Πάρα πολύ σύντομα, παρακαλώ, για να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο και στον Επίτροπο. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε που είστε εδώ. Και λάβατε υπόψη και παρατηρήσεις. Πολύ ενδιαφέρον το έργο σας. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της επιθυμίας για πλούτου και της σοφίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν πάντα εύκολο αυτό. Κοιτάζοντας ε, τώρα όλες τις συμφωνίες που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε, θα καταφέρουμε να σώσουμε το Βιετνάμ από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα λόγω της παραγωγής ε, της ψαρέματος γαρίδας με ένα λανθασμένο σύστημα όχι υγιεινό και πώς αντιμετωπίζει κανείς τα προβλήματα αυτά τα προβλήματα ηθικής φύσης που αφορούν την αλληλεία. Πώς απαντάτε εσείς σε αυτό και με ποιον θα ε, επικοινωνήσετε, με κάποιον για, για τα ε, κοινωνικά δικαιώματα, για να μας δώσετε την κυρία Έλνορ Όστρομ. Η Έλνορ Όστρομ έλαβε το βραβείο Νόμπελ για τα όσα έγραψε σε σχέση με τη διακυβέρνηση των κοινών περιουσιακών στοιχείων, των κοινών αγαθών, των κοινών πόρων. Θα σας πρότεινα να το διαβάσετε. Κύριε Τόμας, για ένα λεπτό κατά ανώτατο όριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη είπαν οι συνάδελφοι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να υπάρχει με την κατάσταση και των, ε, της ε, αλίας και να έχουμε μεγάλες αγωγές. Όχι γιατί καταναλώνουμε στην Ευρώπη περισσότερο ψέρι, αλλά δηλαδή διότι πολύ συχνά οι τιμές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όταν γίνονται εισαγωγές αλλιευμάτων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ζητούμε να καταβάλουν οι αλίες μας και οι παράκτητες περιοχές μας πολύ μεγάλες προσπάθειες και υπάρχουν νόμιμες απαιτήσει, αν θέλετε, όσον αφορά την ανανέωση του αλλιευτικών ε, πόρων και του περιβάλλοντος και ξέρουμε όμως ότι αυτές οι απαιτήσει θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αμοιβαιότητα. Δεν θα μπορούσαμε σε όλες τις συμφωνίες, τις διμερή που έχουμε να απαιτήσουμε να, έχουν, να υπάρχει συστηματικά και ένα κεφάλαιο για την αλία, ώστε μέσω αυτών των εμπορικών συμφωνιών να γίνονται σε όλους γνωστές αυτές οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Πίτροπε. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε εξηγήσω σε τι έγινε τη συνεργασία μας με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ για, αυτό, για όλα αυτά τα ζητήματα, διότι είναι τεχνικά τα ζητήματα που γύρατε και ως επιτοπλίστων θα πρέπει να απευθύνετε τα ερωτήματά σας ε, στην ε, κυρία Δαμανάκη. Η γάμα δέλτα εμπορίου και ως εκ τούτου επίτροπος εμπορίου, υποφαινόμενος, ε, έχει την εντολή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της Ένωσης σε πολύ στενή όμως συνεργασία με τον εκάστοτε επίτροπο, σε συγκεκριμένη περίπτωση με την κυρία Δαμανάκη δεν αποφασίζουμε μόνοι μας επειδή έχουμε τη διαπραγματευτική εντολή, τι παραχωρήσεις θα κάνουμε και τα λοιπά. Ε, ορισμένες φορές χρειάζεται και μία επιδιαιτησία ε, και αφορά αυτό όλους τους επιτρόπους, όχι μόνο την Επίτροπο Αλίας ε, προκειμένου, αλλά και άλλους επιτρόπους Πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον να μην αντιταχθούν σε αυτά που διαπραγματευόμαστε και αποφασίζουμε στη συνέχεια. Δεν είμαι κανένας αγιατολά που αποφασίζω μόνος μου τι πρέπει να κάνουμε στις ε, διεθνείς συμφωνίες. Η Μαρία ούτε καν αυτό θα ήθελε να κάνω. Δεν θα χρειαζόταν να έρχεται και στο Κοινοβούλιο, άμα ήταν έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ένας μόνο τομέας όπου ε, ο εμπλεκόμενος ε, Επίτροπο διαπραγματεύεται μόνος, ε, πρόκειται για τη γεωργία και δεν είναι καλή λύση, Σα το λεω ευθεω ευθέως. Αποφασίστηκε 12-14 χρόνια πριν και ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις διότι προσπαθούν τσακώνονται οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους ακριβώς για αυτό το λόγο. Με τη Μαρία Δαμανέκη δεν είχαμε ποτέ διαφωνίες για οποιοδήποτε ζήτημα μέχρι στιγμής και δεν πιστεύω ότι θα προκύψουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Πρέπει να καταλάβετε το εξής. Ε, η μεγαλύτερη δυσκολία έγινε στο να ε, πείσουμε τους εταίρους μας ότι δεν πρόκειται για και καλυμμένο προστατευτισμό όταν ε, προωθούμε προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε μία από τις συμφωνίες που αναφέραμε με την Νότιο Κορέα που είναι μια σημαντική δύναμη, αλληλευτική δύναμη, ε, επιτυγχάνουμε ε, πολύ καλά αποτελέσματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη όταν οι εταίροι αντιλαμβάνονται ότι είναι και προς δικό τους ε, συμφέρον να πάρουν στα σοβαρά τις ανησυχίες μας για την ευημερία των πολιτών τους. Στις εμπορικές διαπραγματεύσεις λοιπόν που κάνουμε υπάρχει πάντοτε ένα κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα. Και η Αλία είναι ένα τμήμα αυτού του κεφαλαίου. Αυτή τη στιγμή ε, διαπραγματευόμαστε συμφωνία με την ε, Μολδαβία. Είναι περίκλειστη η χώρα και δεν ε, είναι σημαντικός ο κλάδος. Περίκλειστη είναι, τι να κάνουμε. και υπάρχει ο Δνίστερος ε, που είναι το μεγαλύτερο ποτάμι που έχουν και τότε θα υπήρχαν διαφορές με την υπερδνιστερία. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Κορέα με μια περίκλειστη χώρα. Αυτό είναι το αυτό... Σε αυτό το ήθελα να καταλήξω. για την Ταϊλάνδη, διότι έχει μεγάλη σημασία και σχέση με την Αλία, διότι η Ταϊλάνδη είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς αλλιευμάτων, κυρίως για τον κονσερβοποιημένο τόνο. Αυτή τη στιγμή ε, συνεχίζει η διαδικασία εντοπισμού του πεδίου εφαρμογής. Δηλαδή, προσπαθούμε να συμφωνήσουμε για τα ζητήματα επί των οποίων θα συζητήσουμε. Και... Πρόσφατα άρχισαν οι εσωτερικές διαδικασίες, ούτως ώστε επισήμως να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με κοινό στόχο να δρομολογήσουμε τις διαπραγματεύσεις κατά το πρώτο ήμιση του 2013 εξασφαλίζοντας ε, ταυτόχρονα ότι ένα από τα ζητήματα θα είναι ε, τα λιευτικά. Ένα από τα ερωτήματα της κυρίας Φράγα θα ήθελα να σχολιάσω τώρα για τις επιπτώσεις τέτοιου είδου συμφωνιών για την Παπουασία Νέα Γουινέα παραδείγματος χάρη. Είναι προφανές ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιπτώσεις διότι ε, έχει ε, καθολικά διαφορετικό τρόπο ε, για τα λιεύματα της ε, η χώρα, δηλαδή μπορούν σκάφη άλλων κρατών να εκφορτώσουν στην Παπουασία Νέα Γουινέα τα λιεύματα για να κονσερβοποιηθούν. Πρέπει να ε, το λάβουμε αυτό υπόψη όταν συνυπολογίζουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας τέτοιας συμφωνίας. δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, διότι η θάλασσα Bismarck που ε, συνορεύει, που βρέχει την Παπουασία Νέα Γουινέα είναι ένα από ε, μία από τις βασικότερες περιοχές αλίευσης ε, του τόνου. Δεν ξέρω, ο Μπίσμαρκ ποτέ δεν πήγε εκεί και δεν ξέρω γιατί ονόμασαν τα ύδατα με το όνομά του, αλλά είναι πολύ πλούσια αλίευτική περιοχή και με στη συμφωνία με τη χώρα αυτή προέκυψαν ζητήματα με βιομηχανίε και εργοστάσια που ε, φύτρωσαν σαν τα μανιτάρια μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ε, κυρία Λέβιν, ε, μου μιλήσατε για μια ταινία σχετικά με την κονσερβοποίηση του τόνου στην Παπουασία Νέα Γουινέα. Μάλλον πρέπει να διαβάσουμε και το βιβλίο αυτό που προτείνατε εσείς. Κύριε Τόρνβαλντ. Να σας πω τι ξέρω για αυτό το θέμα. Πρόκειται ε, για μια έκθεση εξωτερικού ε, εμπειρογνώμονα και ενός άλλου ε, ε και μια άλλη μελέτη που ζήτησε και χρηματοδότησε το Κοινοβούλιο, βάσει τη οποία η συμφωνία IPA έχει τέτοιε επιπτώσει. Ο Ντέβιντ Μάρτιν, εισηγητή τη έκθεση αυτή, και αναφέρει συγκεκριμένα ότι συνολικά επιτόπου θετικά ήταν τα αποτελέσματα της συμφωνίας, δηλαδή ε, θέσεις απασχόλησης για χιλιάδες ε, γυναίκες, δηλαδή ε, συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά τα εργοστάσια είναι γυναίκες. Δεν είναι κακό να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης στην Παπασία Νέα Γουινέα. Έχω πάει προσωπικά εκεί. Και σίγουρα ένα από τα πράγματα που χρειάζονται είναι δουλειές. Ε, δεν έχω δει την ταινία στην οποία αναφερθήκατε. Αλλά το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη του ε, τις μελέτες που ζητά και χρηματοδοτεί το ίδιο και όχι να αμφισβητεί τα αποτελέσματα των μελετών του. Then uh, the question uh, ε, ε, νέες διαπραγματεύσεις τώρα ε, στον Ειρηνικό Οι χώρες με τις περιοχές επιχαίρουν για τις συμφωνίες τα ζητήματα για την αλληλεία. Οι χώρες του ειρηνικού ζητούν επέκταση της ε, ε, εξαίρεσης για τα ε, κατεψυγμένα προϊόντα και θέλουν να μας δώσουν πρόσβαση μέσω διμεριών συμφωνιών με αντιστάθμιση, κάποια δέσμευση από πλευρά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη αλίευση. Αυτά είναι τα ζητήματα επιτάπητος και πρέπει να τα εξετάσουμε περαιτέρω, είναι προφανές. Ε, δεν ε, έχουμε καμία πρόθεση σε άλλες ε, συμφωνίες ή άλλες IPAs να εισαγάγουμε τέτοια ρήτρα σε σχέση με πρόσβαση, δυνατότητα μάλλον εκφόρτωσης αλλιευμάτων ε, άλλων χωρών στην εν λόγω χώρα, το περίφημο Universal Sourcing ο κανόνας προέλευσης έχει ζητηθεί γιατί αφορά σκάφη που δεν έχουν απαραίτητο ε, την σημαία της χώρας, αυτό σχετίζεται και με τους κανόνες που ισχύουν στα μεταποιητικά τους εργοστάσια. Ε, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα τα καταφέρουμε, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να είναι καθολική η πρόσβαση για όλα τα σκάφη ως προς την εκφόρτωση των προϊόντων. Κύριε Γκάλαχερ, ε, θέσατε διάφορα ζητήματα στην παρέμβασή σας και πιστεύω ότι στο, σε μεγάλο βαθμό είναι θέματα αρμοδιότητας ε, της κυρίας ε, Δαμανάκη. Ε, βεβαίως είναι σημαντικό διότι αυξάνεται η πίεση λόγω των εξελίξεων στα άγρια είδη και και θα ε, κάνουμε μια συνολική αποτίμηση της ε, κατάστασης. Ε, δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο. Κανονισμό κανονισμός τώρα για την παράνομη άναρχη και λαθρή αλία. Ε, ακούστηκαν επικρίσεις ότι δεν εφαρμόζεται ε, ταχαίως. Ναι, πρόσφατα έδωσε τα αποτελέσματα. 15 Νοεμβρίου του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε το Πελή στην καμπότη τη Γουινέα, τη Στριλάνκα το, και άλλες ε, χώρες ε, ότι δεν ε, κάνουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση της άναρχης παράνομης και αλαθρέας αλίας. Δεν συνεπάγεται αυτή η απόφαση επιβολή κύρωσης. Είναι το τελευταίο βήμα πριν από την επιβολή κυρώσεων. Δίνεται χρόνο σε αυτές τις χώρες να διορθώσουν ε, ε, τα σχέδιά τους. Ε, αφήστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει σχέδιο δράση για κάθε μία από αυτές τις χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παρακολουθούμε στενά το ζήτημα. Uh, η, περίπτωση της ε, Κορέας, ε, ναι, στα πλαίσια του κανονισμού για την παράνομη ανέργεια και λαθρέα αλία διερευνάται η υπόθεση τώρα, αλλά δεν μπορώ σε αυτό το στάδιο να σχολιάσω περαιτέρω αυτό το ζήτημα. Όταν συζητούμε για την αλληλεία στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών, ε, εμπλέκονται παραδοσιακά τα εξή σημεία. Πρώτον, πρόσβαση στην αγορά. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριου προσδιορίζει ε, το σχέδιο απολευθέρωση για τα λευτικά προϊόντα της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ ε, και οι περισσότερες δασμολογικές γραμμές ε, δεν χαρακτηρίζονται ευαίσθητες ακριβώς διότι εισάγουμε αλλιεύματα που εκπροσωπούν το 65% της κατανάλωσής μας. Έχουμε κάποιες ευαισθησίες για τον κονσερβοποιημένο τόνο, σαρδέλες, ε, σουρίμι και ατζούγες. Ε, επόμενο θέμα, κανόνες προέλευσης. Ε, είναι ε, και τα δυσχερέστερα σημεία συνήθως των διαπραγματεύσεών μας, ε, διότι συστηματικά χρησιμοποιείται το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, αλλά είναι περιοριστικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αλλιεύονται τα ψάρια από τα σκάφη της χώρας εταίρου και αυτό το θέμα αφορά κυρίως τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπου η οικονομία οικονομικοί φορείς ε, δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες επενδύσει για τα λευτικά του σκάφη. Τρίτο σημείο, η βιώσιμη ανάπτυξη. Επ' αυτού επιδιώκουμε οι εταίροι μας να δεσμευτούν και να εφαρμόσουν τα φυσιολογικά διεθνή πρότυπα για την βιώσιμη αλία βάσει της ε, σύμβασης, παραδείγματος χάρη για τα επικαλυπτόμενα ε, είδη, για τα μέτρα του κράτους λιμένα και το καθεξής. Ε, σε μεμονωμένη βάση ενδέχεται να ανακύψουν και άλλα ζητήματα όπως με τον Καναδά παραδείγματο χάρη που διαπραγματευθήκαμε ενισχυμένη πρόσβαση στα λιμάνια ε, του Καναδά καθώς και άρση εξαγωγικών περιορισμών για αλλιευτικά προϊόντα ε, κάποιων επαρχιών. Μία τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω διότι η η ανταγωνισμού και η προστασία των αλληλευτικών μεταποιητικών βιομηχανιών και τα συμφέροντα του κλάδου έχουν ε, αναφερθεί πολλά και στις παρεμβάσεις σας. συμφωνώ, αλλά ε, σκεφτείτε και το εξή. Αν εισάγεται κατά 65% αυτά που καταναλώνουμε και το 35% είναι εγχώριο παραγωγή, ο βαθμός στον οποίο προστατεύεται την εγχώρια παραγωγή δίνει ένα πλεονέκτημα και στους εισαγωγείς. Πρέπει να κάνετε ε, από οικονομικής πλευράς και αυτόν τον υπολογισμό, διότι ο βαθμός προστασίας της οικίας βιομηχανίας ε, της ε, αλληλευτικής ε, βιομηχανίας γενικότερα είναι συνάρτηση της τιμής παραγωγής που ορίζετε εσείς. Ε, δίνει δηλαδή μεγαλύτερο περιθώριο εισοδήματος, περιθώριο κέρδους και άρα γίνεται ένα παζάρι. Και το ζητούμενο είναι η ισορροπία, η οποία όμως αλλάζει από είδος σε είδος. Το να πει κάποιος ότι όχι, εμεί ε, προστατεύουμε την εγχώρια παραγωγή, τελεία. Όχι, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό από οικονομική σκοπιά. Ε, δεύτερον, μας επιτίθενται αγρίως για κάποιες επιδοτήσεις ε, που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή τη παρέμβασή μου σα μίλησα για την Τόχα. Και ένα από τα ζητήματα που πάντοτε ανακύπτει στις διαπραγματεύσεις όταν, για, όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, της LDC, ε, τίθεται το ζήτημα τι θα κάνετε με τις επιδοτήσεις σας για τα σκάφη σας, για τον ντίζελ παραδείγματο χάρη που και ναι. Δεν μπορείτε μονομένα να τα τα πράγματα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επιθετικά συμφέροντα και μας ζητούν κατάργηση των επιδοτήσεών μας. Είναι ευρύτατο το θέμα. και σημαντικό για τα συμφέροντα της Ένωσης. Παρακαλώ να το συνυπολογίζετε και αυτό, αλλά όχι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά είναι ε, κομμάτια μιας ε, μεγαλύτερης ε, εικόνας. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε, διότι παρά τις υποχρεώσεις σας είσαστε εδώ. Πρέπει να σας επαναλάβω και πάλι ότι είναι ανοιχτή η πόρτα μας. Όποτε θέλετε και για οποιοδήποτε θέμα είστε καλόδεχτες εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως θα μπορούσε να απαντήσει κάποιες από τις ερωτήσεις που έκανα η Επιτροπή, παρακαλώ. Ακόμη και σύντομα. Αναφερθήκατε μόνο σε μένα λέγοντας τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να μου πείτε κάτι και για τον ΠΟΕ. Ίσως αν δεν έχετε την απάντηση στην ερώτηση που έκανα, μπορείτε αργότερα να μου την κοινοποιήσετε. But, uh, Ναι, υπάρχει μια εκκρεμούσα υπόθεση ενώπιον του ΠΟΕ και αυτό που κάναμε εμείς από πλευράς ε, Γενικής Διεθνής Εμπορίου είναι ότι προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε εκτός των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Το αντιμετωπίζουμε ως μια ανεξάρτητη υπόθεση ενώπιον του ΠΟΕ. Φυσικά υπερασπιζόμαστε την υπόθεσή μας, αλλά θα Πρέπει να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης. Ο Καναδάς και η Νορβηγία επίσης έχουν αυτή την υπόθεση ενώπιον του ΠΟΕ. Αλλά δεν το αναμειγνύουμε αυτό με την εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Δεν έχει τίποτα να κάνει με την αλληλεία. Και αν θέλετε να προσφύγετε στον ΠΟΕ μπορείτε. Μας είπαμε, αλλά δεν θα τα αναμίξουμε με τις διαπραγματεύσει ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά. Το ίδιο συμβαίνει και για τις φώκες. Ε, uh, Απαντάει αυτό την ερώτησή σα. Uh, ναι, είναι καλή απάντηση πολιτική, αλλά εγώ ζήτησα ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και αυτό που λέτε βέβαια ότι δεν το αναμεγνύετε, ίσω να μην είναι αρμοδιότητά σα, κύριε Επίτροπε. Απλά πείτε μου το. Αλλά εγώ αναρωτιόμουν ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και κατά πόσο σα ζητήθηκε να εκφράσετε απόψει σε σχέση με τι θέσει του Καναδά και τη Νορβηγία και σε σχέση με τι φώκε. Επίτροπο, όπω σα είπα, μόλι, κύριε Γκάλαχερ, έχουν ε, επανυποβάλει την υπόθεση. Υπάρχει μια καθιερωμένη διαδικασία βάσει της οποίας ε, πρέπει να απαντήσει κανείς μια σειρά ερωτήσεις και μετά μια ομάδα θα αποφασίσει για την υπόθεση και μπορεί κάποιος να κάνει και έφεση στο αποτέλεσμα της διαδικασίας ε, και η όλη διαδικασία χρειάζεται περίπου δύο χρόνια ξέρετε απλά το απομονώσαμε αυτό από τις διαπραγματεύσεις διότι είναι σαφές ε, ότι δεν πρόκειται να επιληθεί στο πλαίσιο το χρονικό των διαπραγματεύσεων έχει μόλις ξεκινήσει ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτό το πρόβλημα είναι να λυθεί μια απόφαση από τον ΠΟΕ. Και στη συνέχεια το κάθε μέρο ε, ένδικο μέρο να ε, πράξει ανάλογα βάσει αυτής της απόφασης αλλά ε, δεν θα επιληθεί πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και τα δύο μέρη θεωρούν ότι δεν έχουν δυνατότητα συμβιβασμού. Είναι πολύ σαφές, οπότε το διατηρήσαμε εκτός των διαπραγματεύσεων. Πολύ εντάξει. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Επίτροπο. Τώρα ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων για το πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής και Μαυριτανίας. Προσωρινά λοιπόν φεύγω από το Προεδρείο για να σας παρουσιάσω το θέμα αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Okay, ε, Συνάδελφοι, αναλαμβάνω προσωρινά την Προεδρία για να μιλήσουμε για το πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Η συγγετής, ο κύριος Αντροβέρ, του δίνω μέσο το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντω από εδώ μπορώ να μιλήσω πιο ήρεμα για ένα θέμα το οποίο λυπάμαι δυστυχώς που δεν είναι ο κύριος Ντεπιπέρ εδώ. Λέω ότι λυπάμαι διότι στην προηγούμενη συνεδρίαση αυτή τη Επιτροπής μετά από τις εξηγήσει και τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει φαίνεται τουλάχιστον αυτή είχα την εντύπωση ότι, ότι μας είχε πείσει ο κύριο Πιπέρ αλλά φαίνεται ότι το αντίθετο συμβαίνει. Ή δεν καταλάβαμε τίποτα, ή δεν κατάλαβε τίποτα. Διότι ούτε εμένα με έπεισε, ούτε ε, μπορώ να συμφωνήσω. Σήμερα λοιπόν λέω όχι με, για την συμφωνία αυτή. Λέω όχι για αυτή τη συμφωνία, διότι λέω ότι ναι, θέλουμε συμφωνία με τη Μαυριτανία, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικό, αλλά προφανώς όχι αυτή την συμφωνία, διότι είναι αρνητική. Σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε. Δεν έχει μεγάλο νόημα η τελεγή απόψεων, διότι δεν υπάρχει τίποτε το καινούριο. Δεν υπάρχει κανένα καινούριο θέμα που θέλω να αναφέρω στην Επιτροπή. Πρόκειται για ποιο σημαντική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί και, ε, και αυτό αφορά και τα αλλιεύματα και τα αντισταθμίσματα με τον προπολογισμό. Πρέπει να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις εδώ και 15 μήνες διαρκούν για μια διετή συμφωνία, πράγμα που αποδεικνύει όχι μόνο ότι υπάρχει δυσκολία, αλλά και επιπροσθέτως ότι κάτι, κάτι αποτύχαμε. Το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει υπογράψει την προσωρινή του εφαρμογή και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να θέσω και να μου απαντήσουν αν προβλέπετε κάτι τέτοιο να γίνει στο άμεσο μέλλον και είναι αληθές ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορώ να πω ότι έχει μόνο αρνητικά σημεία, κάτι θετικό θα έχει. Θεωρητικά δίδει ε, προτεραιότητα πρόσβασης στον αλλιευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα δοθούν σε άλλους αλλοδαπούς ε, στόλους ε, προτεραιότητα και προνόμια που δεν θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πολύ σημαντικό επίση το θέμα της στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή εδώ έχουμε να κάνουμε με οκτώ κατηγορίες που αφορούν διαφορετικές δραστηριότητες και με σημαντικά αντισταθμίμασματα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Η έκθεσή μου, ε, στην έκθεσή μου θα έχω πάρα πολλά επιχειρήματα και υπέρ του ναι και υπέρ του όχι. Πάρα πολύ σημαντικά επιχειρήματα. Θα τα επαναλάβω πολύ συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα, όπως έχω πει πολλές φορές και κάθε μέρα είμαι και πιο πεπισμένος, αυτή η συμφωνία έγινε χωρί να ληφθεί υπόψη ούτε ο επαγγελματικό κλάδο, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κλάδο Ελίας είπε πριν από την 6η, 7η, 8η συνάντηση με την Επιτροπή, δεν ξέρω πόσε συναντήσει έγιναν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όταν ήδη όλοι ξέραμε ότι στην 5η είχαν κλείσει τα περισσότερα θέματα και έτσι το κατανοώ δεν είχε την ε, σαφή εικόνα του τι ακριβώς γίνεται. Πρέπει να πω ότι όλα έγιναν πίσω από την πλάτη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του τομέα, διότι και εμείς δεν μπορέσαμε να γνωμοδοτήσουμε για την ε, συμφωνία αυτή. Είναι λοιπόν εντελώς αρνητική, διότι δεν επιτρέπει την πρόσβαση του δικού μας στόλου, που είναι, αποτελείται από 32 σκάφη, 24 τα οποία είναι ισπανικά. Πρέπει να πω ότι απερχαιωμένες εκθέσεις ελήφθησαν υπόψη για να γίνει συμφωνία, οι πολύ πιο πρόσφατες στις οποίες λέγεται ότι δεν χρειάζεται να περιοριστεί ή να απαγορευτεί η πρόσβαση αυτού του ελευτικού στόλου δεν ελήφθη υπόψη. Ελέχθη καταρχάς ότι δεν υπήρχαν δυνατότητες αλίες και μετά ψηλοάλλαξαν τα πράγματα λέγοντας ότι τον αλληλευτικό στόλο το δικό της ήθελε να χρησιμοποιήσει μόνο η Μαυριτανία. Τώρα, για τα πελαγικά είδη. Ε, βλέπουμε ότι έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αλλιευμάτων. Πράγμα το οποίο είναι πολύ κακό και για την ευρωπαϊκή περίπτωση και για τους ίδιους τους πλειοκτήτες. Πράγμα που σημαίνει ότι για αυτούς το κόστο ανεβαίνει σε ποσοστό 300 με 400%. Και αν δούμε και τα έμεσο κόστος το οποίο ε, υπάρχει το ότι θα πρέπει 60% να, ε, οι ναύτες να είναι από τη Μαυριτανία. Ποιο είναι το συμπληρωματικό κόστος από τη μεταφορά. Και όλα αυτά τα θέματα μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι απαράδεκτες οι συνθήκες που προβλέπονται για τον ολευτικό στόλο από οικονομικής πλευράς και ου μόνον. Και βεβαίως δεν θα μιλήσω για τις ζημίες που υφίστανται και τα λιμάνια. Εμένα, πόσο με αφορά, τα δύο λιμάνια των Καναρίων, Δελαλούθ και ε, Λαπάλμα. Πιστεύω δηλαδή ότι παρά το γεγονό ότι μα είπε πάρα πολλέ φορέ η Κομισιόν ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη από όλε τι δυνατέ συμφωνίε που θα μπορούσε να συνάψει, για μένα είναι μια συμφωνία που δεν τη θέλει ο τομέα των επαγγελματιών του Δεν τη θέλει ο κλάδο των επαγγελματιών. Δύο ερωτήσει θέλω να κάνω στην Κομισιό σε σχέση με δύο διαφορετικά θέματα, αλλά έχουν σχέση μεταξύ του. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να μου πει με σαφήνεια, γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να μου πει, πόσα σκάφη χρησιμοποίησαν τι ε, ε, άδειες που έχουν δοθεί από τότε ε, που υπεγράφει η συμφωνία. Πιστεύω κανένα ο, πόσα ε, από σκάφη που ε, ψαρεύουν πελαγικά είδη, πόσα από αυτά τα οποία ε, ψαρεύουν ψαρεύουν οστρακοειδή. Για να μου πει και ανάλογα με τον αριθμό θα δούμε για ποιους λόγους γίνεται ό,τι γίνεται. Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί αρκετά είναι ότι όπως παρατηρήσαμε σε μια πολύ πρόσφατη συνεδρίαση σε επίπεδο Κορεπέρ, ότι άλλαξε η νομική βάση στη συμφωνία και από όπως πάντα να έχουμε το 43-2 άρθρο λέμε τώρα το άρθρο 43 συν τίποτε άλλο σαν να λέμε η συνθήκη χωρίς να λέμε ποιο άρθρο θα ήθελα να εξηγηθούν ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή και δεύτερον θα ήθελα να μου πει ποια είναι η θέση της Επιτροπής σε σχέση με αυτή την αλλαγή. Δηλαδή αν συμφωνεί, αν δεν συμφωνεί και αν δεν συμφωνεί τι θα κάνει ή τι σκέφτεται να κάνει για αυτή την αλλαγή την οποία εμείς δεν την καταλαβαίνουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν την καταλαβαίνω. Και θα ήθελα να μου πείτε γιατί έγινε ότι έγινε. Θα κάνει κάτι η Επιτροπή. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προσφύγουμε κατά της απόφασης αυτής. Θα ήθελα λοιπόν από πρώτο χέρι να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Βεβαίως, ε, αν μου ζητήσετε, έχω και άλλα στοιχεία να σας δώσω. Πρέπει να σας πω ότι ως εισηγητού η θέση μου θα είναι σαφέστατη. Να μην ε, υπογράψουμε την συμφωνία αυτή, να μην την επικυρώσουμε, διότι ούτε εμείς την επιθυμούμε, ούτε ο κλάδος και θα πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Όχι μόνο όταν, όχι αφού τεθεί σε ισχύ, όπως προτίθεται η Επιτροπή, διότι όπως προβλέπετε, προβλέπονται τέσσερις μήνες για να ε, φανεί αν είναι χρήσιμη μια συμφωνία ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι ήδη με το ότι να είναι όλοι αρνητικοί και να μην χρησιμοποιούν ε, τα ενδεχόμενα ωφέλη της, όλοι απέδειξαν ότι δεν του αρέσει. Έχουμε λοιπόν αυτή την δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων μηνών, πράγμα το οποίο είναι παράλογο, διότι προβλέπει πώς θα χρησιμοποιηθεί στους τέσσερις μήνε, αλλά από τη στιγμή όμως που εφαρμόζεται προσωρινά και επικυρώνεται, οι πληρωμές για κάποιες ποσότητε θα πρέπει να γίνουν στο τρίμηνο. Άμα λοιπόν πληρωθούν στην Μαυριτανία τα 70 ε, δις, πώς θα μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω. Διότι ξέρουμε από τις προηγούμενες επιτροπές ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. Έχω λοιπόν πάρα πολλά επιχειρήματα για να πω όχι σε αυτή τη συμφωνία. Ναι όμως για να ψάξουμε ε, μία καλύτερη συμφωνία με καλύτερες, καλύτερους όρους και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Μαυριτανία. Εδώ δεν θέλουμε να κερδίσει ο και να χάσει ο άλλος. Θέλουμε η συμφωνία να είναι θετική και να βγουν κερδισμένοι όλοι οι εταίροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σάντζες Πεσέρο, Ιζαμπέλα Λεβίν, Μιράντα Πατράου no. Ναι. είναι στη, στον κατάλογο των ε, ομιλητών. Κύριος Πρεσέδο, ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ούτε θα επαναλάβω τα επιχειρήματα του εισηγητού του κ. Μάτο. Γενικά, συμφωνώ απόλυτα, αλλά θα πρέπει να πω ότι την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι σήμερα δεν βλέπω να υπάρχει λόγος για να αλλάξω τη σχέση μου ή για να αμβλυνθούν οι ανησυχίες μου. Όντω είπαμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η συμφωνία αυτή με την Μαυριτανία. Το μόνο που θα πω είναι ότι εδώ και κάποιο καιρό έκανα μία ερώτηση προς την Κομισιό, λέγοντας για ποιο λόγο ε, ο αλλιευτικός στόλος των κεφαλοπόδων που ψάρευε τα κεφαλόποδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απομακρύνθηκε από την ε, Μαυριτανία. Εγώ πήρα την ε, έκθεση, την ε, σχέδιο συμφωνίας, τη διάβασα, αλλά τα πράγματα είναι χειρότερα. Τώρα, με τα θέματα της ε, βιομάζας, μεταξύ άλλων επίσης προβλέπονται αλλαγές. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πρώτα απ' όλα, από όσο ξέρω, δεν θα πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες, αλλά θα πρέπει να μειωθεί πράγμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκλειστεί ο αλευτικός στόλος της Ευρώπης, αλλά ίσως ε, μείωση του αριθμού των σκαφών. Δεύτερον, αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτή την έκθεση είναι ότι έχει 900 μικρά λευτικά σκάφη η Μαυριτανία, κανό άλλα μικρά και 200 άλλα ε, σκάφη ε, ξένα τα οποία έχουν ε, πάρει αυτή τη στιγμή σημαία μαυριτανική. Θα ήθελα να ξέρω, η δική μας, συγγνώμη, θα ήθελα να ξέρω τώρα αυτά τα σκάφη τα οποία πήρανε τώρα την ε, νέα σημαία της Βρυτανίας θα πρέπει να αλλιεύουν τα κεφαλόποδα. Επίσης, οι πληροφορίες που προέρχονται από τον κλάδο και από το Ινστιτούτο το Ισπανικό της Οκεανογραφίας αναφέρουν ότι όλο και περισσότερο ε, αυξάνονται τα αλλιεύματα σε μία τελευταία συνεδρίαση με εκπροσώπους της κυβέρνησης και εκπροσώπων την ε, ε, σε Μαυριτανίας ε, αναφερότανε ότι βάσει κάποιων ιδιωτικών συμφωνιών ε, υπήρχαν πάρα πολλά ε, κινέζικα αλλιευτικά σκάφη με σειρώμενα δίκαια, τα οποία, δίχτυα τα οποία αλλιεύαν. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι έχουμε αποκλεισμό για να μπορέσουν να αλλιεύσουν τα δικά μας σκάφη τα κεφαλόποδα, πηγαίνουν ξένα και κάνουν τα ίδια πράγματα. Βλέπω λοιπόν ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια να είναι κατά κάποιο τρόπο εξισορροπημένη η συμφωνία αυτή και καμία προσπάθεια να καταβάλλεται και εκ μέρους της Μαυριτανίας. Δηλαδή, οι αλλιευτικοί ε, πόροι αυτή τη στιγμή είναι με τον αποκλεισμό του αλευτικού τόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάθεση και των μαυριτανικών ε, σκαφών και των άλλων αλλοδαπών από τρίτες χώρες. Όλο και περισσότερο λοιπόν αυξάνονται οι ανησυχίες μου. Εγώ έκανα, υπέβαλα ερώτηση στην Κομισιόν για όλα αυτά τα θέματα, καμία απάντηση δεν πήρα. Πιστεύω ότι έχει μεγάλες ανισορροπίες αυτή η συμφωνία και θα δημιουργήσει προηγούμενο και θα αποδυναμώσει την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις μετέπειτα συμφωνίες που θα μπορούσαν ε, να συναυθούν στον τομέα αυτό, μειώνονται πολύ και περιορίζονται τα δικαιώματα αλίευσης, προβλέπονται κάποιες πρακτικές οι οποίες έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιες περιοχές και θα έπρεπε να απαγορευτούν και διαρωτώ με και θα ήθελα να μου απαντήσει η Κομισιόν εάν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ε, κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε τους πόρους που υπάρχουν. Ε, αν μπορεί κάποιος να μου πει κάτι, να μου το πει, διότι αυτή τη στιγμή έχω ανησυχίες και βλέπω ότι είναι αρνητική αυτή η συμφωνία και δεν νομίζω ότι μπορεί να την υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η Ισαμπέλα Λέβιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από μερικά χρόνια, το 2011 νομίζω το 2010, αυτή η Επιτροπή έστειλε μια ανταπροσωπεία στη Μαυριτανία με την κυρία Φράγκο, τον κύριο Φερέρα, εμένα και άλλους και συναντηθήκαμε με εκπρόσωπους του τομέα στη Μαυριτανία κατέστη πολύ σαφές εκείνη τη στιγμή ότι τα κεφαλόποδα τα ήθελαν για τη δική τους βιομηχανία. Είχαν αλληλευτικές δραστηριότητες κεφαλόποδων, ήθελαν να τα αναπτύξουν, είχαν μηχανότρατες και ήταν ένα που ήθελαν να αναπτύξουν σε ένα κοινό ψήφισμα που υπέγραψαν το ΕΛ και οι σοσιαλιστές, το ΑΛΔΕ, οι πράσινοι και η ΓΚΟΕ στις 10 Μαΐου 2011 το παρόν κοινοβούλιο δήλωσε ότι ε, επειδή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Μαυρετανία βοήθησε στην εκμετάλλευση ορισμένων αποθεμάτων όπως το, ε, τα χταπόδια έδωσε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη σε επιχορηγούμενα τέλη για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου το Μάιο του 2011. Υπογραφική από όλες τις ομάδες. Επίσης αναφέρει ότι η, η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει συμμόρφωση με τις βιώσιμες αλίες, ειδικότερα όσον αφορά τις συστάσεις χορήγησης ε, προτιμησιακής πρόσβασης σε πόρους σε τοπικούς αλληλεί στη Μαυριτανία. Αυτή ήταν λοιπόν η βούληση αυτού του κοινοβουλίου που αποτέλεσε εντολή του Κοινοβουλίου προς την Κομισιόν για να πάει να διαπραγματευτεί μια νέα αληθική συμφωνία με τη Μαυριτανία. Ακούγοντα κάποιο τη συζήτηση σε αυτή την επιτροπή, δημιουργεί την εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο ήταν κατά. Αλλά ουσιαστικά μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ. Κοιτώντας μετά το τι λέει το Συμβούλιο, το Συμβούλιο λέει στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2012 ότι, λόγω, ότι στην εξωτερική πολιτική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οι προτεραιότητες των παρακτών κρατών υπέρ των δικών τους ελευθερικών τομέων. Τι θέλει λοιπόν ο ελευθερικός τομέας της Μαυριτανίας, εδώ έχω μια έκθεση και σύσταση από την κοινωνία των πολιτών της Μαυριτανίας, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην ΟΑΞΟΤ τον Οκτώβριο του 2012, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι οργανισμοί αλλιέων της Μαυριτανίας. Μπορείτε όλοι να διαβάσετε αυτή την έκθεση. Υποστηρίζουν ισχυρά αυτό το πρωτόκολλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι για πρώτη φορά έχουμε μια δίκαιη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επικροτούν και θέλουν όλες οι άλλες αλληλευτικές συμφωνίες που συνάπτει η μαυριτανική κυβέρνηση με άλλα ξένα αλληλευτικά κράτη να έχουν σχεδιαστεί βάσει του της ίδιας αυτής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε την πρωτοπορία της στον τομέα της βιωσιμότητας μιας ξένης χώρας ε, που δραστηριοποιείται στην Αλία. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε. Ουσιαστικά την περασμένη εβδομάδα όταν ψηφίσαμε όλη την εκθεσή μου για την εξωτερική διάσταση της κοινής ελευθερικής πολιτικής, όλες αυτές οι αρχές ε, επιβεβαιώθηκαν ξανά μια μεγάλη πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου θεωρεί ότι η προτιμησιακή πρόσβαση πρέπει να δοθεί σε παράκτια χώρα. Είναι φυσικό. Δεν πιστεύω ότι κανείς ε, Ισπανός παραπονιέται αυτή τη στιγμή για τα κεφαλόποδα. Αν σας έλεγε κάποιος επιστήμονας από τη Μαυριτανία ότι υπήρχε περίσευμα κεφαλόποδων στα νερά της Γαλλικίας και οι αλληλείς ε, της Γαλλικίας θα ήθελαν πρόσβαση εκεί. Θα αφήνατε τους Μαυριτανούς να έρθουν να τα ψαρέψουν διότι υπάρχει περίσσια. Η Μαυριτανία είναι μια ανεξάρτητη χώρα και αν η Μαυριτανία θέλει να διατηρήσει τους δικούς της αλληλευτικού πόρους εκεί πρέπει να το κάνει και πρέπει να το αποδεχτείτε. Επίσης πρέπει να αποδεχτείτε ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών του Συμβουλίου και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου πιστεύουν ότι αυτές οι αρχές κυριαρχούν επί των πάντων και ότι οι, επιχειρήσεις, οι ελευτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα για αυτά τα συμφωνίε πρόσβαση. Την περασμένη εβδομάδα το ψηφίσαμε ότι πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ελευτική Βιομηχανία πρέπει να ε, επιφορτίζεται με ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους όταν έχει πρόσβαση σε ξένα ύδατα στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνίες. Το ψηφίσαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα. Πέρυσι ψηφίσαμε επίσης το ίδιο ακριβώς πράγμα και επίσης και το Συμβούλιο έχει την ίδια άποψη. Λέει ότι το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του λέει ότι χωριώντας εξουσιοδοτήσεις αλληλείας μέσω τελών που πληρώνουν οι διοκτήτε Ευρωπαίοι για τις αλληλευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι δίκαιες και αντίστοιχες στα ωφέλη που παρέχουν οι συνθήκες πρόσβασης. Αυτή είναι η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να το δεχτείτε. Εάν οι αλληλευτικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν είναι επικερδείς αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να επιχορηγούμε μη βιώσιμη αλληλεία μέσω συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να εξαναγκάζουμε τρίτες χώρες να πουλάνε τους ελληνικούς τους πόρους εάν δεν το επιθυμούν. Ευχαριστώ. Thank you, Isabella. Uh, the next is... Ευχαριστούμε, Ιζαμπέλα. Άννα Μιράντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, cualquiera de nosotros que estamos aquí somos de... Εμείς εδώ είμαστε Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές. Δεν είμαστε ευρωβουλευτές τη της Μαυριτανίας είτε άλλες χώρες. Είμαστε ευρωβουλευτές. Κάποιοι έχουν ε, συμφέροντα τις εκλογικές τους επιχειρήσεις στους πολίτες τους. Εγώ θέλω να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα όσων κάνουν αηφόρο αλληλεία. όπου και να την κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, ή στην Ισπανία ή στην Μαυριτανία. Και βεβαίως τα οικονομικά αντισταθμίσματα δεν νομίζω ότι μπορούν ε, να δώσουν κάτι σε αυτούς οι οποίοι κάνουν ερασιτεχνική αηφόρο λίγη. Επίσης θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε και τον βαθμό της διαφθοράς. Τώρα, εάν πρόκειται για μία σωστή έκθεση, θα την υπερψηφίσω. Πιστεύω ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου είναι ε, Αν είναι δίκαια αυτή η συμφωνία, συγγνώμη, και το αποφασίσει το κοινοβούλιο θα την ψηφίσω. Αλλά δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Όπω είπε και ο πρόεδρο, πρόκειται για μια συμφωνία που για πέντε μήνε άφησε την ε, αλληλεία ε, στη μοίρα τη, δεδομένου ότι έγιναν διάφορες αλλαγέ για τη νέα συμφωνία βάσει απερχαιωμένων και παλιών εκθέσεων. Ξέρουμε ότι θα υπάρχει και ε, οικονομικό βάρος για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη. Έλεγε η Επίτροπος ότι δεδομένου ότι είναι παράδοξη αυτή η κατάσταση ή δεδομένου ότι υπάρχουν προβλήματα δεν θα συνεχίσουν ε, να δραστηριοποιούνται τα κοινοτικά λευτικά σκάφη. Εμείς δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε με οποιοδήποτε τίμημα και περισσότερο από τα, τους Μαυριτανούς, τους δικούς μας Θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία που δεν είναι αυθαίρετη και που να είναι δίκαιη. Αν πρόκειται για συμφωνία η οποία έκλεισε διότι υπάρχουν ε, ε, σφάλματα και λάθη που ελήφθησαν υπόψη, έχω αμφιβολίες. Θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή Ποιες είναι οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των ε, ευκαιριών που προσφέρονται για αλεία. Φαίνεται ότι είναι πολύ μικρά τα ποσοστά. Α μου πει η Κομισιόν. Και δεν είναι και παρόν και το Συμβούλιο σήμερα. Τι θα γίνει αύριο στο Συμβούλιο, θα υπάρξει μειοψηφία που θα μπλοκάρει ψηφοφορία, θα υπάρξει μειοψηφία, διότι αυτή τη στιγμή αν μπλοκαριστεί αυτό το πρωτόκολλο που έχει προσωρινή ε, εφαρμογή, τι είδου ε, οικονομικά ε, προβλήματα θα υπάρχουν. Και τι κάνουμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Όμοιροι είμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Ενώ ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις τελικά. Διότι ήδη υπάρχει αυτή η προσωρινή συμφωνία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εδώ και πέντε μήνες υπάρχουν άτομα που περιμένουν να ε, τους επιτραπεί να δραστηριοποιηθούν στο Μοράγκο, στο Καρί, σε άλλες μέρες της Γαλλικίας, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία που να τους το επιτρέπουν για να τους επιβεβαιώνουν κάποια πράγματα. Και σε ένδειξη αλληλεγγύης θα πω το εξή. Αυτά τα λευτικά σκάφη είναι αυτά πρέπει να πληρώσουν ε, ε, διότι έγιναν κακά οι διαπραγματεύσει. Η κυρία Γαρθία Γέρμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα συγκρίνω το πρωτόκολλο αυτό με το προηγούμενο, που δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω το πρωτόκολλο με τη Βοζανβίκη και ήμουν και εγώ εισηγήτρια και την ε, μελέτησα και βεβαίως ε, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος Αντώνη Σάντσες Πρεσέδο. Υπάρχει όμως, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θέλω να αναφέρω, άλλες ανησυχίες τις οποίες θέλω να εκφράσω και που δεν ελέγξαμε. Πρώτο θέμα, πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε καλή συμφωνία που να είναι συμφανή με αυτή την ε, πρόσβαση προτεραιότητας ε, στην ε, Μαυριτανία. Μιλώ για τον κοινοτικό ε, αλλιευτικό στόλο. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα εδώ. Παρά όταν έχουμε ένα πιο δημοκρατικό και ανοιχτό πολίτευμα σε άλλες χώρες. Γίνονται επικρίσεις, αναφέρεται ότι είναι κακή η συμφωνία αυτή, κακό το πρωτόκολλο και όπως είπα, κάνοντας σύγκριση με το πρωτόκολλο της Μοζαμβίκης, τα ποσά τα οποία δίδονται για να υποστηριχτούν οι δραστηριότητες των αλλιέων στην ε, Μαυριτανία. Τρία εκατομμύρια είναι ένα ελάχιστο ποσό. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε από τα 70 εκατομμύρια ή μπορούμε να προσφέρουμε κάτι πιο γενναιόδωρο εμείς οι Ευρωπαίοι που όχι μόνο πηγαίνουμε εκεί για να αλλιεύσουμε αυτό το οποίο ως προϊόν και το θέλουμε για να το καταναλώσουμε και είναι μια οικονομική ε, δραστηριότητα που μας αποφέρει, αλλά το αφαιρούμε και από τα άτομα τα οποία ενδεχομένως θα το στερηθούν. Τώρα, όταν γίνεται λόγος για συμβάσεις με τους ναυτικούς, προβλέπεται σύμφωνα με τη ρήτρα ότι οι ναυτικοί, τα πληρώματα των ε, αλληλευτικών στόλων θα είναι κατά 60% Μαυρίτανοι. Διαφορετικά θα πρέπει να πληρώνετε ένα ποσό για καθέναν. Τι κάνουμε λοιπόν. Κάνουμε εμείς μία συλλογική σύμβαση. Θέλουμε να δώσουμε εγγύηση στους εργαζομένους. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε όχι μόνο για να βοηθήσουμε τους εργοδότες και τον τομέα, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε και τον εργαζόμενο. Αυτό δεν το βλέπω εδώ. Στη Μοζαμβίκη έλεγε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να ε, προσληφθούν δύο ε, ναυτικοί. Ενώ εδώ γίνεται λόγος για κάποιους ναυτικούς οι οποίοι θα πρέπει να είναι από την χώρα της σημαίας και αναφέρονται και κάποια δικαιώματα ε, για τους εργαζόμενους, αλλά υπό τις συνθήκες που επικρατούν και θέλουν να επιβάλλουν οι Μαυριτανοί. Πιστεύω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Ξέρω ότι σιγά σιγά περικόπτονται πάρα πολλά δικαιώματα και μετά πληρώνουμε τις επιπτώσεις, έτσι. Διότι αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση κρίσης που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίο. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι ότι τα μέτρα ελέγχου δεδομένου ότι είπαμε ότι θα υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή τους ε, καθημερινή. Τα μέτρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να βελτιωθούν. Προς δικό μας συμφέρον. Οι Ισπανοί θέλουμε όλες αυτές ε, οι φέζες ζώνες που υπάρχουν όσον αφορά ε, την Ισπανία, τη χώρα μου να σταματήσουν να υπάρχουν. Θα ήθελα να γίνει κάτι σωστό και οι μελέτες επιπτώσεων θα πρέπει να επιτρέπουν όταν υπάρχουν αμφιβολίες ή εμφανίζονται κάποιες λανθασμένες ιδέες για τους Ισπανούς πριν να βγουν προς τα έξω, να κάνει κάποιος αντιπαραβολή με τα πραγματικά στοιχεία. Εδώ γίνεται λόγος ε, για ποσοστά ειδών διατροφής που θα δώσει κανείς στους Μαυριτανούς 2% των πλεονασμάτων. Ακούστε, είπαμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό. Είμαστε Ευρωπαίοι. Δεν είμαστε ούτε από τις Κανάριες, ούτε από τη Μεσόγειο, ούτε από τη Μαδρίτη, ούτε από τη Γαλλικία. Εμείς είμαστε με το σύνολο του κλάδου, με το σύνολο των αλλιέων. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει το μοντέλο ανάπτυξη να είναι και κάπως ανθρωποκεντρικό, διότι δεν το κάνουν όλοι αυτό και δεν το προβλέπουν. Ευχαριστώ. Επόμενο στη λίστα είναι η κυρία Μπιλμπάου. Κύριε Τσάσκουν Μπιλμπάου, ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω κάποια από τα επιχειρήματα τα οποία άκουσα στις παρεμβάσεις των συναδέλφων αλλά θα ήθελα η Επιτροπή να απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο στις εξής ερωτήσεις που θα γίνουν. Πώς χρησιμοποιήθηκαν οι άδειε που δόθηκαν από τον τομέα αυτό μέχρι σήμερα, εάν δεν χρησιμοποιήθηκαν, ποια είναι η δική σας αξιολόγηση του γεγονότος αυτού, για αυτή, γιατί εάν δεν υπάρχει συμφωνία εκ μέρους του ε, ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εσείς θέλετε να υπάρξει αλλαγή της νομικής βάσης παρά το ότι διαφωνεί το Κοινοβούλιο. Ποιες είναι οι αιτίες για τις οποίες όντως βγάλατε από τη συμφωνία τα κεφαλόποδα για επιστημονικούς λόγους έγινε κάτι τέτοιο. Βάσει ποιων επιστημονικών εκθέσεων και εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι, αν οι ίδιοι οι Μαυριτανοί, οι αλληλείς, ο κλάδος, η κυβέρνηση της Μαυριτανίας δεν το ήθελε. Ε, τι ακριβώς συμβαίνει. Δώστε μας συγκεκριμένες απαντήσεις. Και τελικά, θα ήθελα να πω ότι το να επιβάλλει κανείς στον τομέα αυτό μια συμφωνία με την οποία όλος ο κλάδος διαφωνεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι με άλλες ιδιωτικές συμφωνίες ξένοι στόλοι αλλιεύουν αυτά τα, αυτούς τους πόλους, ποια είναι η πόρους, ποια είναι η στρατηγική της Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι αν πρέπει να έχουμε τον ηγετικό ρόλο όσον αφορά την ε, αηφόρο αλληλεία, την προστασία του περιβάλλοντος και όλες τις άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε υιοθετήσει και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε το καλό παράδειγμα, ακόμη και σε διεθνές επίπεδα, θα ήθελα να μου απαντήσει η Κομισιό, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη, ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει μελλοντικά. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε με μία συμφωνία από την οποία έφυγαν τα κεφαλόποδα. Υπάρχουν άλλα αλλιευτικά σκάφη εκεί με ε, σημαία της Μαυριτανίας που ψαρεύουν αυτά τα είδη. Και ποια θα είναι, επαναλαμβάνω, η στρατηγική σας στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα και με τις άδειες και ο τομέας ε, επειδή είναι αντίθετο δεν έχει ζητήσει ούτε μία μοναδική άδεια. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια έκθεση που δεν θα χρησιμοποιηθεί, διότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ενισχύει την εικόνα μας. Και εάν κάνουμε κάτι τέτοιο, το μόνο που θα κάνουμε είναι να κατασπαταλήσουμε πόρους και χρόνο. Πόρους γενικότερα σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό παρακαλώ την Κομισιό να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν σήμερα εδώ, ώστε όλοι και όλοι λες να μπορούμε να κάνουμε την κατάλληλη αξιολόγηση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η επόμενη στον κατάλογο είναι η Κάρμεν Φράγκα. Δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά θέλω να κάνω κάποια σχόλια έχοντας ακούσει συναδέλφους. Εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο εγκρίθηκε ένα ψήφισμα, αλλά είναι επίση αληθές ότι αλλάζουν τα πράγματα. Και αν όντω το ψήφισμα αυτό για τα κεφαλόποδα βασίστηκε σε μία μελέτη του 2008, είναι αληθές και το ξέρουμε όλοι ότι εκ των υστέρων έγινε και μία περαιτέρω μελέτη από, η κάποια, από κάποιο οικιανογραφικό Ινστιτούτο και η κατάσταση ήταν εντελώ διαφορετική. Ακούστε τώρα. Η Μαυριτανία μπορεί να απαντήσει, να αποφασίσει ότι ό,τι είναι καλύτερο ως αλίευμα το θέλει για τον εαυτό της, το δικό της ε, αλευτικό στόλο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εποφελές για τον ε, ε, μικρό αλιέα. Θα επωφεληθεί από όλη αυτή την κατάσταση ο στόλος, ο κινέζικος με άλλη σημαία. Άρα όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία εντελώς λαθασμένη έτσι όπως παρουσιάζεται. Λοιπόν, ένα από τα κυρία θέματα για κάποιος στα πλαίσια του ψηφίσματος είναι στις επόμενες διαπραγματεύσεις να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες αλίας βάσει των κατάλληλων τεχνικών μέσων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πέτυχε εδώ και είναι μία από τις αδυναμίες στην παρούσα ε, Σωστά το λέει και η κυρία Λέβιν. Άμα δεν θέλει αλλού δύο συμφωνία με Βρυτανία, α μην κάνει. Δικό τη κυρίαρχο δικαίωμα είναι. Αλλά αν ε, Παρά το γεγονός λοιπόν ότι όλος ο αλλιευτικός στόλος και όλοι οι παρόντες από τη δίκηση είπαν ότι δεν θέλουν να υπογραφεί η συμφωνία, πώς το υπέγραψε, θέλει να το υπογράψει η Επιτροπή. Αλλά σε τι χρησιμεύει μια εμπορική συμφωνία που δεν έχει καμία χρησιμότητα. Επίσης, ελέγχθη από κάποιον ότι οι αλληλείς και όλος ο κλάδος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εγώ μπορώ να σας πω ότι Δεδομένου ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια δημοκρατική χώρα, πολλοί δεν μπορούν να πούνε κουβέντα. Και πρέπει να πω ότι πάρα πολλοί στα διάφορα λιμάνια της χώρας αυτής περνάνε πάρα πολύ άσχημα, έχουν χάσει τη θέση απασχόλησή τους και θέλουν να έχουν ένα μηνιαίο μισθό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό γίνεται στο λιμάνι του Εμπαλού από τότε που δεν μπορεί να αλλιεύσει ο κοινοτικό στόλο. Ευχαριστώ. Η Μαρία Πατραονέβες. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ούτε εγώ είχα την πρόθεση να παρέμβω και μου, εφόσον μου δώσατε όμως ε, το λόγο, παρότι αρνήθηκα, ακούγοντας ε, παρεμβάσεις όπως αυτήν της Κάρμεν ένιωσα την ανάγκη να παρέμβω κι εγώ. Θα είμαι σύντομη γιατί είναι τόσο απλό αυτό το ζήτημα για μένα. Είναι τόσο παράλογα απλό το ζήτημα που πραγματικά αναρωτιέμαι για τι πράγματα μιλάμε. Και θα ήθελα να μ' ακούσει η Ιζαμπέλα Λέβιν, ε, γιατί διαφωνώ μαζί τη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα ότι θα είμαι σύντομη γιατί είναι πάρα πολύ ε, και ε, απλό το ζήτημα και παράλογα απλό. Πρέπει να είναι υποφελή συμφωνία και για τους δύο συμβαλωμένους. Δεν, είναι, δεν εξυπακούεται αυτό και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μέρος που είναι ικανοποιημένο και το οποίο υπερασπιζόμαστε γιατί τα είπαμε εδώ, η συμβαστική μας λύση εδώ είναι καλή για τον ευρωπαϊκό στόλο. Και πολλές φορές το ξεχνούν αυτό κάποιοι. Οπότε δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Εάν δεν θέλει τη συμφωνία ο στόλο, εμείς θα κάνουμε. Θα επιβάλλουμε τη συμφωνία σε κάποιον ε, ενώ δεν τη θέλει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Οι περικοπές που έγιναν για ε, τα κεφαλόποδα που θέλουν ε, οι Ισπανοί, μα και οι Πορτογάλοι τα θέλουν. Αυτά δεν το καταλαβαίνω υπάρχουν ε, συμφέροντα τμήματων του ευρωπαϊκού στόλου που δεν κατοχυρώνονται, ε, κατοχυρώνονται συγγνώμη, Υπάρχουν όλα αυτά τα ε, ε, οικονομικά ζητηρήματα ε, υπερβολικά περίπλοκα, μα δεν είναι καλή συμφωνία γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν. Έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα και επαναλαμβάνω, η, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δεν δίνουμε χρήματα σε κάποια χώρα για οποιοδήποτε λόγους που παρεπιπτόντως δεν καταλαβαίνω ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε καμία συμφωνία πρέπει να είναι αμοιβαίω επωφελή η συμφωνία και αυτό το λόγο είναι απλό για να πρέπει να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω Σας ευχαριστούμε Τώρα θα ακούσουμε τον Μάρκ ε, Τζόνσον. Εσείς υποθέτω θα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσετε τουλάχιστον να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Θα βάλω τα δυνατά μου για να απαντήσω και θα, σίγουρα θα προσπαθήσω να απαντήσω τα συγκεκριμένα ερωτήματα που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτού το κάνω αυτό και με τον κίνδυνο να επαναλάβω αυτά που είπαν ε, οι συνάδελφοι πριν από τρεις εβδομάδες, ε, σχολιάζοντας κάποιες πτυχές ε, της συμφωνίας, θα πρέπει παρόλα αυτά να επανέλθω σε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Για μας είναι ξεκάθαρο στην Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι είναι η βέλτιστη δυνατή συμφωνία, διαθέσιμη συμφωνία αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε καλύτερη συμφωνία και οπωσδήποτε θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Όταν δηλαδή εξετάζουμε ε, τις επιπτώσεις της άρνησης χορήγησης εγκατάθεσης από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μάτο είπε ότι συνεχίζει, μπορεί να συνεχιστεί η αλίευση. Μάλιστα, αληθεύει αυτό. Βάσει του άρθρου 9 της, ε, του κανονισμού περί αδειοδότησης ε, για την αλλιεύση. όμως αυτό περιορίζεται σε ένα εξάμεινο μετά την εκπνοή του προηγούμενου πρωτόκολλου και αυτό εξέπνευσε τον Ιούλιο του 2012. Αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει η ώρα για την αλία δύο μήνες έχουμε ακόμη για δύο μήνες έχουν οι στόλοι που θέλουν να αλλιεύσουν να αλλιεύσουν. Όταν τώρα παρέλθουν και αυτοί οι δύο μήνες και αποφασιστεί να μην δοθεί σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, τότε θα υποχρεωθούμε να στείλουμε κοινοποίηση στη Μαυριτανία ότι δεν θα επικυρωθεί η συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σταματήσει η αλίευση και ε, θα επανέλθουμε για να διαπραγματευτούμε νέα συμφωνία. Και αναφέρθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τη μορφή μιας μελλοντική συμφωνίας ε, και το χρόνο ε, που χρειαζόμαστε για να διαπραγματευτούμε μια κακή συμφωνία. Εγώ θα αναρωτηθώ το αντίστροφο. Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να διαπραγματευτούμε μια καλή συμφωνία. Όχι ψευδεστήσεις παρακαλώ. Δεν θα υπάρξει καμία αλίευση για πολύ καιρό αν δεν ανανεωθεί το πρωτόκολλο. Λοιπόν, για τα δύο συμβαλόμενα μέρη και το αν είναι αμοιβαίω επωφελή συμφωνία, γιατί αυτό απασχόλησε πολλού από του ομιλητέ. Θα πρέπει να επανέλθω ε, για τα κεφαλόποδα. Θα πρέπει να επανέλθουμε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων των συμφωνιών. Λοιπόν, διέπονται από την σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αυτές τις συμφωνίες και είναι ξεκάθαρο ότι Βάσει αυτών των συμφωνιών αυτό που χορηγείται στις τρίτες χώρες είναι το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα δεν ορίζεται από την τρίτη χώρα αλλά από τη χώρα που έχει το πλεόνασμα. Ε, μπορούμε εμείς να αλλιεύσουμε το πλεόνασμα σε ύδατα τρίτης χώρας. Εάν η τρίτη χώρα επιθυμεί να αλλιεύσει ολόκληρο το απόθεμά της για να αναπτύξει περαιτέρω το στόλο της, έχει δικαίωμα και ε, ε, συνάδει αυτό απολύτω με το διεθνές ε, δίκαιο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτό το ζήτημα. Πρώτον, το είχαμε στη διάθεσή μας, η απάντηση είναι όχι. Οι Μαυριτανοί δεν δεν θέλησαν να μας δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και ε, ε, να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει άλλος τόλος που να αλλιεύει κεφαλόποδα στη Μαυριτανία. Υπάρχουν κάποια σκάφη που ονομάζουμε εμείς ε, κινέζικα, που... αλλά το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τα ευρωπαϊκά σκάφη, τα χρησιμοποιούν άλλες σημαίες και πάνε και αλλιεύουν σε άλλα διεθνή ύδατα. Έτσι είναι τα πράγματα όμως και το πρώτο εμπόδιο που χρειάστηκε να υπερπηδήσουμε είναι να μας δώσουν τη δυνατότητα οι Μαυριτανοί και δεν έγινε αυτό. Δεύτερον, επιστημονικά τεκμήρια. Εμεί βασιστήκαμε στα επιστημονικά στοιχεία της Οικονομικής ε, και ε, Τεχνικής και Επιστημονικής Επιτροπής, όπως κάνουμε πάντοτε. Η ΣΤΕΑΦΚ μας δίνει τα στοιχεία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε βεβαίως. Ε, υπάρχει αυτή η μελέτη του Οκεανογραφικού Ινστιτούτου και αναφερθήκατε σε αυτή. Ενδιαφέρουσα είναι και ε, περιέχει διάφορε συστάσεις που ενδεχομένω να οδηγήσουν σε αύξηση του αποθέματο ε, στα μαυριτανικά ύδατα, αν και όταν συμβεί αυτό, αν και όταν η Μαυριτανία αποφασίσουν ορίσουν ότι έχουν πλεόνασμα και δεν ε, θα το αλεύσουν με το στόλο τους και μας το διαθέσουν, τότε δυνάμει του ε, πρωτοκόλλου, γιατί έχουμε μηδενική ποσόστοση για τα κεφαλόποδα, το, το τονίζω αυτό, είναι μηδενική ποσόστοση, οπότε αν αλλάξει αυτό με το νέο πρωτόκολλο, τότε μπορούμε να επανέλθουμε και να διαπιστώσουμε αν έχουμε πρόσβαση ή όχι σε αυτό το απόθεμα. Υπήρξαν και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για την αδειοδότηση και για την ε, χορήγηση αδειών. Όλες οι άδειες για τα αθηνοειδή έχουν ε, κατανεμηθεί, 20 περίπου, ε, και το ίδιο και για την Πολάκα. Για τα πελαγικά δεν έχουν ζητηθεί Καναδίες ε, και ε, εκπλησόμαστε πραγματικά διότι πλησιάζει η εποχή αλίευσης, ε, ούτε και για τις γαρίδες. αλλά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο από βιολογικής πλευράς είναι περίοδος ανάπαυλας, οπότε αυτό δεν μας ξαφνιάζει. Ε, θα αναφερθώ τώρα στο θέμα της νομικής βάσης. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η Επιτροπή πρότεινε τρία ε, μέσα. Ε, το ε, πρώτο προτάθηκε βάσει του άρθρου 43 εδάφιο 2 της Συνθήκης Λιταργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με το 218 εδάφιο 6 της ίδιας συνθήκης. Αυτό το μέσο απαιτεί σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και βάσει αυτού συνάπτεται η συμφωνία. Έγιναν συζητήσεις στο Συμβούλιο ε, και πιστεύω ότι το είναι δουλειά του Συμβουλίου να ε, μιλήσει για τα πεπραγμένα. Πάντως, σε βάση του άρθρου 43, εμεί μένουμε στη θέση μας ότι δηλαδή το άρθρο 43 εδάφιο 2 είναι η πρόσφορη νομική βάση και δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε τη θέση μας σε σχέση με αυτό ως προς την κατάσταση για την προσωρινή εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Ε, είπαμε ότι έχουμε αυτό το παραθυράκι. Δύο μήνες υπολείπονται και βάσει των τελευταίων συμφωνιών, ε, ε πληροφοριών που διαθέτουμε το Συμβούλιο την Δευτέρα που μας έρχεται θα εγκρίνει την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας. Δηλαδή δεν θα βασιζόμαστε στον κανονισμό για τις αδειοδοτήσεις αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε την αλίευση επί τη βάση του πρωτοκόλλου. Με την διάμεση εφαρμογή τότε θα συνειδητοποιήσουμε ε, πόσες άδειες θα χορηγηθούν βάσει του πρωτοκόλλου και τότε θα συζητήσουμε με τους Μαυριτανούς ε, για ε, ενδεχόμενες προσαρμογές των διατάξεων περιαδιών μέσα στο πρωτόκολλο και έχουν δείξει ένα σχετικό άνοιγμα οι μαυριτανικές αρχές για αυτό το ζήτημα. Βεβαίως αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο ξαναλέω του ισχύοντος πρωτοκόλλου. για τις υπόλοιπες ε, αλληλευτικές δυνατότητες που ε, τέθησαν στη διάθεσή μας ανάμεσα στο υφιστάμενο και το προηγούμενο πρωτόκολλο, δηλαδή δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές. Τα κεφαλόποδα είναι η μοναδική εξαίρεση και αληθεύει ότι τροποποιήθηκαν οι τεχνικοί όροι, οι οποίοι όμως ε, προσδιορίζονται βάσει περιβαλλοντικών ανησυχιών και επιχειρημάτων που σχετίζονται με τη διατήρηση του αποθέματος.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 Ε, για την κλαδική στήριξη. 3 ε, εκατομμύρια από τα 17. Λοιπόν, η κλαδική στήριξη, η στήριξη του κλάδου θα πρέπει να ερμηνευτεί διαφορετικά. Βάσει του προηγούμενου πρωτόκολλου ήταν ε, πολύ πιο περιορισμένη υποστήριξη. Δεν έχει όμως απορροφηθεί πλήρως το κονδύλι και τα νέα κονδύλια δεν μπορούν να εκταμιευθούν μέχρι να απορροφηθούν τα προηγούμενα και γινόμαστε σε ένα επίπεδο που αντιστοιχεί στην ικανότητα απορρόφησης ε, και στις ανάγκες, στις τωρινές ανάγκες της Μαυριτανίας ε, σε σχέση με την απέτηση να έχουμε ναυτικούς μαυριτανούς εν πλώ. Όντως ε, ζημιώθηκε αύξηση και πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς συμφέρον και των δύο μερών, αλλά ως προς τους μισθούς ε, που ε, πληρώνονται δεν ε, υπήρξε αύξηση, καμία αλλαγή και στο προηγούμενο πρωτόκολλο αναφέρεται ότι καμία διαφορά δεν υπάρχει ανάμεσα στο προηγούμενο που εξέπνευσε την 1η Ιουλίου που σας είπα και το νέο που διαπραγματευόμαστε τώρα. Για να κλείσω και την παρέμβασή μου. Θα έλεγα ότι ευελπιστούμε σε μια ταχύ εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας ε, και τα σκάφη που ακόμη δεν έχουν ε, λάβει άδειε, ε, θα τις λάβουν και θα χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες αλλιευτικές δυνατότητες και στη συνέχεια αν διαπιστώσουμε πρόβλημα σε σχέση με τη χορήγηση αδειών να μην ξεχνούμε ότι υπάρχει μέρη μνήμα μέσα το πρωτόκολλο για αναστολή τετράμινη αν δεν υπάρξει χρήση των διαθέσιμων αδειών. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Κατάλαβα ε, ότι η κυρία Φράγα έχει επερώτηση για ένα από τα δύο ερωτήματα που, στα οποία μόλις απαντήσατε. Παρακαλώ. Ε, Θέλω να πω το εξής. Κύριο εκπρόσωπο τη Επιτροπής είπε ότι έχουμε όλες τις αδειοδοτήσεις για τα θηνοειδή και για και για την Πολάκα. Αλλά νομίζω ότι για τα υπόλοιπα είδη άλλαξαν πάρα πολύ οι συνθήκες και κυρίως για τα κεφαλόποδα και για άλλα πελαγικά είδη. Εδώ επίσης ελέγχθη ότι για και για τα οστρακοειδή ε, υπάρχει κάποια αλλαγή, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι αυτή τη στιγμή κανένα αλλιευτικό σκάφος που αλλιεύει την Πολάκα να μην αναπτύσσει δραστηριότητες στην περιοχή αυτή. Μπορεί να απαντήσει η Κομισιόν. Ε, πιστεύω ότι μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι εμείς έχουμε διαφορετικές πληροφορίες όσον αφορά τη δόση των αδειών και τις ελληνικές δραστηριότητες. Εμείς ξέρουμε ότι οι ελληνικές δραστηριότητες έχουν αυξηθεί και όσον αφορά τον Μαύρο Μερλούκιο ουσιαστικά έχουν αυξηθεί οι ποσότητες ανάμεσα στα δύο πρωτόκολλα. Ναι, ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στον εισηγητή λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω από την Κομισιόν, διότι πραγματικά εγώ εκτιμώ τις προσπάθειες που έγιναν για να υπερασπιστούν αυτά που δεν μπορούν να υπερασπιστούν. Το, η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Για ποιον? Για ποιον? Θα πρέπει να είναι για τον ίδιο τον κλάδο και για τη Μαυριτανία, αλλά και εμείς ε, πρέπει να υπερασπιστούμε το δικό μας ελληνικό στόλο που είπε δεν, τον, δεν τη θέλουμε αυτή τη συμφωνία. Και αν δεν το θέλει αυτό ο λευτικός τόλος και ο κλάδος, γιατί κάνει τέτοια προσπάθεια να επιμένει σε αυτή τη συμφωνία. <coughs> Κυρία Φράγκα ρώτησε, πείτε μας, πόσα είναι τα πλοία τα οποία αφορά αυτή η κατάσταση. Ένα, δύο, τρία, πέντε, εκατό. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, τα καλύτερα για την πελαγική αλία, για όχι... Πείτε μας συγκεκριμένα τι περί πρόκειται. Επίσης, Εάν 15 ε, μήνε χρειάστηκε για να διαπραγματευτούμε μια κακή συμφωνία, πώ θα χρειαστούν για μια καλή. Ή τόσο ή, ή λιγότερους μήνες. Τον ίδιο χρόνο αναλόγουμε. Τέτοιου είδους διαπιστώσεις, τι να πω, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τα κεφαλόπεδα. Οι Μαυριτανοί δεν ήθελαν να μας τα διαθέσουν και τα αλλιευτικά σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνται για αυτή την αλία είναι της Μαυριτανίας. Εντάξει. Αλλά μετά μας λέει η Κομισιό ότι οι επιστημονικές μαρτυρίες λέγουν ότι δεν μπορούν, αλλά δεδομένου ότι αυτό το θεωρούν πολύ θετικό, αν αλλάξει η κατάσταση θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε. Ποια είναι η κατάσταση. Θα αλλάξει η κατάσταση και τι θα σημαίνει αυτό. Ότι θα υπάρχουν περισσότερα αποθέματα ότι άλλαξαν οι επιστημονικές μαρτυρίες και θα έχουμε μία συμπληρωματική άδεια. Ότι τώρα και για έξι μήνες ψαρεύουμε αυτό που θέλουμε εμείς και έξι μήνες θα μοιραστούμε αυτές τις ποσότητες. Επίσης, η νομική βάση. Εμένα πολύ καλό μου φαίνεται αυτό που λέει, δηλαδή ότι θα πρέπει να μας εξηγήσει το Συμβούλιο γιατί την άλλαξε. Εντάξει, η Επιτροπή μας λέει ότι έτσι έχει η νομική βάση ότι θα πρέπει να είναι το 43-2 και δεν θα οπισθοδρομήσει. Η ερώτησή μου είναι σαφέστατη. Τι σημαίνει αυτό. Θα επιτρέψει η Κομισιό να αλλάξει το 43-2 και να υπάρξει ως βάση μόνο το 43 γενικότερα. Επίσης, οι προσωρινές αξιοδιοτήσεις. Από την πρώτη στιγμή μας λέει η Επιτροπή ότι θα πρέπει προσωρινά η δεδότηση να δοθεί το συντομότερο δυνατό για να λειτουργήσει το πρωτόκολλο. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το σχήμα και πόσες άδειες θα δοθούν ε, και μετά θα δούμε. Γιατί δεν το κάνουμε ήδη. Αφού ήδη πέρασαν τέσσερις μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων μπορέσαμε να δούμε πόσες ε, αδειοδοτήσεις ζητήθηκαν. Α, τι άλλαξε. Ας δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται. Ούτως ή άλλως ε, το υπάρχει δυνατότητα να πάρει κάποιο άδεια, αλλά δεν ζήτησε κανένα. Τώρα, ή πρόκειται για προσωρινή εφαρμογή ή όχι, δεν αλλάζει τα πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μπλα μπλα και να πούμε πολλές γενικότητες, αλλά όπως Έλεγε και η Ζαμπέλα, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε και δεν πρέπει σε κανένα να υποχρεώσουμε ε, να μας πουλήσει τους πόρους που διαθέτει αν δεν θέλει. Αλλά κανένας δεν μπορεί να μας υποχρεώσει να αγοράσουμε για κάτι που δεν θέλουμε. Γιατί λοιπόν κάνει τέτοιου είδους ε, προσπάθειες η Κομισιόν. Ε, το ψήφισμα του Μαΐου 2011 πρέπει να πω ότι όπως είπε και η κυρία Φράγκα δεν ισχύει και δόθη εντολή στην Κομισιόν. Και αυτό το οποίο θέλουμε να δοθεί διαφορετική εντολή στην Κομισιόν, δηλαδή να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία. Διότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έγινε. Επίσης, αν η Μαυριτανή κυβέρνηση λένε ότι θα θέλανε όλες οι συμφωνίες ε, να είναι παρεμφερής με την τωρινή. Βεβαίως. Και εμένα, αν μου δίναν πιο πολλά λεφτά ως κυβέρνηση. Αν είναι δικά μου τα πληρώματα. Αν ε, πληρώνω τα καύσιμα, αν μου πληρώνω τα καύσιμα. Τι ωραία. Ευλογημένου είδο συμφωνία είναι αυτή που θέλει να υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα νέο επιχείρημα υπέρ της ε, χορήγησης ε, συμφωνίας για αυτή το πρωτόκολλο, θα ήθελα να παρακαλέ, να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να μην την εγκρίνει αυτή τη συμφωνία, αλλά να την ξαναρχίσει. Καλύτερα τώρα παρά μετά από τέσσερις μήνες που θα έχει καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά και θα έχουμε έναν αριθμό αδειών που κανένας δεν θα έχει ζητήσει να χρησιμοποιήσει και θα έχουμε δημιουργήσει και περαιτέρω δυσκολίε για τον ελληνικό στόλο όλου του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ενδιαφέρουσα την συζήτηση και πιθανώς θα τη συνεχίσουμε σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αλλά προς το παρόν το σημείο αυτό της ε, ημερήσιας διάταξης ε, έχει κλείσει. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και θα συνεχίσετε με άλλον πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Αλλάζω καπελάκι. Παίρνω την θέση και πάλι του Προέδρου και θα μιλήσουμε το επόμενο θέμα, αλλιευτικέ δυνατότητε για την οικονομική αντιπαροχή που προβλέπει η Συμφωνία Αλλιευτική Σύμπραξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου. Θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με εισηγητή τον κύριο Σάντζε Πρεσέδο. Του δίνουμε στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, σήμερα είναι μια ανταλλαγή απόψεων για αυτή τη νέα συμφωνία. Εγώ θα απλώ θα ήθελα να αναγγείλω ότι ήδη έχω κάνει το σχέδιο ε, εκθεσής μου. Η θέση μου είναι θετική. Είμαι θετικός για την, ε, ε, για την έγκριση της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου, αλλά με ενδιαφέρουν και δικές σας απόψεις. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Μαυρικίου άρχισαν το 89 και μέχρι το 2007 συνεχίζονται οι συμφωνίες. Το τελευταίο, το πρώτο ήταν 2003-2007. Από το 2007 δεν έχουμε κανένα νέα, ε, νέο μέσο που να μας επιτρέπει να έχουμε συγκεκριμένη συμφωνία με το Μαυρίκιο και βάσει ιδιωτικών συμφωνιών δραστηριοποιούνταν οι στόλοι, οι διάφοροι. Λοιπόν, η νέα συμφωνία και η το νέο πρωτόκολλο θέλουν να αποκατασταθεί η κατάσταση αυτή και να αναλυφθούν δημόσιες και να γίνει επίσημη συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας του Μαυρικίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες για το τι μπορεί να είναι αφενός η η αλλιευτική αυτή συμφωνία ή η ευρύτερου περιεχομένου η, η οικονομική η μεταξύ Μαυρικίου και Οικονομικής Ένωσης. Προβλέπεται ένα πρωτόκολλο τριετές 60 εκατομμυρίων ευρώ που είναι ποσό μικρότερο από αυτό που προβλέπεται ε, για μία τριετία το σχετικό έγγραφο στρατηγικής ε, του Μαυρικίου για το 2003-2007 προβλέπει για την ε, μακροοικονομική πολιτική 70 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια 12,4 για επίγουσες δράσεις και για συνδρομή άλλου τύπου. Άρα, σφαιρικά στα πλαίσια της οικονομικής ε, βοηθείας και συνεργασίας με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Μαυρίκιο προβλέπονται κονδύλια 2 δις ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για ένα μικρό ποσό. Η δημοκρατία του Μαυρικίου έχει 1.300.000 κατοίκους με εισόδημα ανακεφαλή 15.000 δολάρια έχουν ε, σημαντική αποκλειστική οικονομική ζώνη και κυρίως η Αλευτική Συμφωνία με μας περιλαμβάνει την αλίευση των οειδών 85 αλλιευτικά ε, σκάφη και χίλιους τόνους λιγότερους ε, ε, από ό,τι την προηγούμενη συμφωνία. Εγώ προσπάθησα να μελετήσω αυτή τη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αναφέρεται συμπερασματικά ότι δεν υπάρχουν από οικονομικής πλευράς ή από κοινωνικής πλευράς ή όσον αφορά την προσοχή του περιβάλλοντος αρνητικές επιπτώσεις, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς θα πρέπει να πω ότι ο Μαυρίκιος, σύμφωνα με το έγγραφα στρατηγικής του Μαυρικίου, έτσι όπως ε, αναφέρει η Κομισιό, συμπεριφέρεται καλά όσον αφορά τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα, είναι δημοκρατική χώρα, τηρεί τους κανόνες διαφάνειας και διαβούλευσης και παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι κάποιες οργανώσεις αλλιέων από τον Μαυρίκιο ήρθαν σε επαφή μαζί μου, είπαν ότι δεν ικανοποιούνται, δεν τους ικανοποιεί πάρα πολύ η εξέλιξη όλης αυτής της διαδικασίας. Εγώ έκανα, επέβαλα ερώτηση στην Κομισιό, αλλά ακόμη δεν έλαβα απάντηση. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει να πούμε ότι η διαφάνεια στον τομέα της αλίας είναι ένα από τα θεμελιώδους σημασία θέματα, δεδομένου ότι η αλευτική πόρη είναι μέλος του φυσικού περιβάλλοντος όλων μας, άρα οτιδήποτε γίνεται θα πρέπει να έχει αυτή την δημόσια διάσταση, τον δημόσιο χαρακτήρα, τον ανοιχτό. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να διευκολύνουμε την ύπαρξη ιδιωτικών συμβάσεων και συμφωνιών όσον αφορά αυτούς τους φυσικούς κοινούς πόρους. Βεβαίως ε, δεν είναι συμβατή αυτού του είδους η αλία με την ε, αλία που αφορά τα σαλιευτικούς πόρους παραδοσιακά του Μαυρικίου, δεν χρησιμοποιούνται οι ίδιες τεχνικές, δεν χρησιμοποιούνται οι ίδιοι, ε, τα ίδια αλλιευτικά σκάφη, οι ίδιες τεχνικές και η αλληλεία αφορά κυρίως τα θηνοειδή. Η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής ε, του Ινδικού ωκεανού για τα τονοειδή λέει ότι δεν υπάρχει υπεραλίευση τονοειδών στην περιοχή αυτή, άρα δεν νομίζω ότι ούτε για την αηφορία της αλίας, ούτε για την τοπική αλία δεν υπάρχει κάτι το αρνητικό. Η αλία είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες του πληθυσμού του Μαυρικίου. Υπάρχει όμως ε, πολύ καλή συμπεριφορά εκ μέρους της ε, οικονομίας ε, του νησιού αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξουμε την υπογραφή της συμφωνίας αυτής της νέας και του πρωτοκόλου. Βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση και εκ μέρους του επαγγελματικού κλάδου. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μου και θα ήθελα να μου πείτε και εσείς, συνάδελφοι, ποιοι είναι, ποια είναι η θέση σας. Αν ε, επιτρέπετε η Κομισιόν πρώτα απ' όλα να λάβει το λόγο. Κύριος Τζόνσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η εισηγητής είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας. Είναι σημαντική η συμφωνία αυτή για εμάς, διότι θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε σε ένα σωστό πλαίσιο τη συνεργασία μας. Η συμφωνία αυτή βασίζεται στις αρχές της μεταρρύθμισης. Έχουμε λοιπόν εκεί μέσα όλες τις ρήτρε που θα περίμενε κανείς να δηλαδή, δει σε νέα γενιά συμφωνιών αλληλευτικής σύμπραξης. Θα έλεγα επίσης ότι χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε θέση να αντικαταστήσουμε τις συμφωνίες παλιάς γενιάς του 90 με μια συμφωνία νέα γενιά. Οι συνθήκε, οι όροι τη συμφωνία περιγράφηκαν λεπτομερώ από τον κύριο Συγητή. Όσον αφορά την ερώτηση που θέτει ο κύριο Συγητή σε σχέση με τη διαφάνεια, συμφωνούμε. Η διαφάνεια είναι σημαντική. Εμείς επιχειρήσαμε να τη διασφαλίσουμε πριν από τη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία και μετά τις διαπραγματεύσεις. Ο κ. Συζητητής ε, ανέφερε την εκτίμηση αντικτύπου, την αξιολόγηση που διεξάγαμε. Αυτό έγινε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Είδαμε τι γινόταν στο παρελθόν, τι θα γίνει τώρα και κοιτώντας και προ το μέλλον. Αυτό έγινε με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου, ο οποίος ε, ταξίδεψε στο Μαυρίκιο, ήρθε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους εκεί αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουμε και έναν επιτετραμένο για την αλληλεία, ο οποίος ενεπλάκει επίση σε επαφές με τους ενδιαφερομένους και κατά το 2011 έλαβαν χώρα τρεις διαφορετικέ συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους και το 2012 έλαβε χώρα μια άλλη σειρά συναντήσεων με τους ενδιαφερομένους για να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, Πώ δηλαδή θα λειτουργεί πρακτικά αυτή η συμφωνία. Ένα άλλο σημείο που σχετίζεται με τη διαφάνεια είναι ότι όταν η κοινή επιτροπή συνεδριάζει, τα πρακτικά δημοσιεύονται δημόσια. Αυτό έχει προβλεφθεί. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα της διαφάνειας και πιστεύω ότι αυτή η πρακτική είναι καλή και θα μπορούσε να αναπραχθεί και αλλού. Ευχαριστώ κυρία Λέβεν. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα μπορούσα να μην επικρίνω αυτή τη συμφωνία, αλλά μου κάνει έκπληξη που και ο εισηγητής και η Κομισιόν μιλάνε για τα υψηλά επίπεδα διαφάνειας αυτής της συμφωνίας και ότι όλοι οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι έδωσαν την άποψή τους και ότι όλοι συμφωνούν με αυτή τη συμφωνία διότι μου έφτασαν πληροφορίες από την κοινωνία των πολιτών του Μαυρικίου όπου είναι ιδιαίτερα αναστατωμένοι επειδή δεν συμμετείχαν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Έγιναν ε, συνεδριάσεις, ε, συναντήσεις με άλλη συνδικάτα, την Αλληλευτική Ένωση, διότι γνωρίζετε είναι μεγάλος τουριστικός προορισμός ε, και έχουν και πολύ μεγάλες εταιρείες ψυχαγωγικής αλληλείας καθώς και οι ενώσει καταδύσεων αντέδρασαν έντονα διότι δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Είναι ιδιαίτερα αναστατωμένοι λόγω της έλλειψης διαφάνειας τη διαπραγματεύτική διαδικασία και ότι, από το γεγονό ότι δεν ενημερώθηκαν καταλήλως δυστυχώ από τη δική τους κυβέρνηση και ότι το μόνο που άκουσαν, το μόνο που έμαθαν ε, ήταν η δημοσίευση του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο φέτος. Επίσης είναι δυσαρεστημένη με τη χαμηλή χρηματική ανταμοιβή που λαμβάνει ο Μαυρίκαιος. Ένα κιλό τόνου αξίζει 6,5 ευρώ, δηλαδή 2,6 ρουπίες Μαυριτανίας και στην αγορά όπου εκφορτώνονται τα ψάρια, τα λεύματα στο Μαυρίκιο, η τιμή του τόνου είναι 90 ευρωπίες το κιλό. Πιστεύουν λοιπόν ότι ουσιαστικά χαρίζονται οι πόροι. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη της Κομισιόν και του κυρίου Σιγητή. Έχετε ακούσει τίποτα για αυτά τα παράπονα και ποιες είναι οι απόψεις για αυτά. Επίσης θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους τα διάφορα ψηφίσματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει όλοι όπου λέμε ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει και σε τρίτες χώρες και ότι η διαφάνεια πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες. Αυτή είναι λοιπόν μία μου ερώτηση. η μία μου ερώτηση. Μια άλλη ερώτηση είναι ότι αν εδώ μιλάμε, αν εδώ πρόκειται για συμφωνίες νέας γενιάς, αναρωτιέμαι για το άρθρο 11, το οποίο μου είναι πρωτόγνωρο. Δε, υπό την επικεφαλίδα εμπιστευτικότητα αυτό είναι ένα νέο άρθρο. Εμπιστευτικότητα δεν υπήρχε στα παλιά πρωτόκολλα, στι παλιέ συμφωνίε, όπου διασφαλίζεται ότι όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αγλευτικές δραστηριότητες θα θεωρούνται εμπιστευτικά. Και αυτό μου έκανε έκπληξη. Δεν είναι ακριβώ αυτό που περιμέναμε ούτε αυτό που περίμεναν οι πολίτε του Μαυρική. Θέλουν να ξέρουν πόσα σκάφη βρίσκονται εκεί και τι αλλιεύουν. Σκόπιμο θα ήταν αυτέ οι πληροφορίε να είναι δημόσιε. Επίση, ανησυχώ επίση για την έλλειψη περιφερειακή προσέγγιση σε αυτή την περίπτωση, διότι έχουμε και τη συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη, την οποία ετοιμάζουμε και τη συμφωνία με τι Κομόρες ένα από τα καλά πράγματα με το πρωτόκολλο της Μαδαγασκάρης είναι ότι συμπεριλαμβάνει τους καρχαρίες ως ε, ιδιαίτερο τμήμα όχι απλά ως τα αλλιεύματα για την αλληλεία τόνου αλλά και με ειδικέ ποσοστώσεις και εδώ αυτό δεν το βλέπω ερώτηση μου λοιπόν προς την Κομισιόν είναι γιατί δεν κοιτάξετε το πρωτόκολλο με τη Μαδαγασκάρη Υποθέτω ότι μιλάμε για παρόμοιο τύπο αλίας με παρόμοιο τύπο παρεπιπτόντων των αλλιευμάτων. Ορισμένα από αυτά τα παρεπιπτόντα αλλιεύματα βρίσκονται σε ε, επικίνδυνη θέση και ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Τέλος, ε, θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα σε σχέση με τη χρηματική συμβόλη των πλειοκτητών. Αυξήθηκε σε τι επίπεδο βρίσκεται σε σχέση με άλλα πρωτόκολλα, το πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία για παράδειγμα. Δεν βρίσκω λεπτομέρειες ε, γι' αυτό στη συμφωνία. Θα ήθελα να μου πείτε δηλαδή πόσο θα πληρώσουν οι πλειοκτήτες εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει, ας ακούσουμε την, ε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις mentioned the, the transparency which we have tried to pursue in relation to this agreement. Um, of course, one σε σχέση με τη διαφάνεια, είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Πάντοτε μπορεί κάποιο να κάνει περισσότερα για τη διαφάνεια. Ε, γυράσκουμε ή διδασκόμενοι και ε, διαβουλεύτηκα με τους εμπλεκόμενους φορείς ε, το 2011. Επανειλημμένα τους ενημέρωσα ε, μετά ε, την συμφωνία θέλουμε να είμαστε διαφανείς και για την εφαρμογή της ε, συμφωνίας θα μπορούσαμε να ανοίξουμε περισσότερο τα δίχτυα μας ενδεχομένως και να ψαρέψουμε και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον και αυτό με φαίνει στο άρθρο 11 για την εμπιστευτικότητα. Το θέμα της εμπιστευτικότητας ε, δεν έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να σταματήσει την κυκλοφορία των πληροφοριών ως αυτό σκοπό. Δηλαδή, ο στόχος είναι η ταυτότητα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτή τη συμφωνία να μην δημοσιεύεται, να μην είναι κοινή γνώση όλων. Υπάρχει και μια δεύτερη αράδα που μιλάει για την ε, χρήση των ε, προσωπικών δεδομένων ε, και πότε προβλέπετε. Ένα λεπτάκι να σας πω και ποιο άρθρο είναι. Σε σχέση με τους καρχαρίες, όντως δεν αναφέρθηκε το ζήτημα σε αυτό το πρωτόκολλο. Σίγουρα θα μας απασχολήσει στο μέλλον και μάλιστα ε, σε σχέση με αυτό το θέμα και τη συμπερίληψη Συμφωνία της Μαδαγασκάρης ήταν χρονικό το ζήτημα. Αλλά θα το έχουμε κατά νου για το μέλλον. Δεν ε, είχαμε αρκετό χρόνο για να συμπεριλάβουμε και αυτό στη Συμφωνία. Αυτό είναι όλο. Ε, σε σχέση τα ποσά ε, της συμφωνίας. Ε, ε, τα ίδια έχουμε για τους πλειοκτήτες, για τις άδειε, όπως και για τα άκρος, όπως και συμφωνίες για τα άκρος μεταναστευτικά είδη. 100 ευρώ ο τόνος, τα 65 από τον προπολογισμό της Ένωσης και τα 35 από το, τα κονδύλια των πλειοκτητών. Ε, ας επιστρέψω στο άρθρο 11. Στη δεύτερη πρόταση λέει ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την, ε, τους σκοπούς της εφαρμογής της συμφωνίας ε, και για το σκοπό διαχείρισης παρακολούθησης ε, ελέγχου των αλλιευμάτων συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές δηλαδή. Λέμε ότι όντω ναι, τα δεδομένα για τους πλειοκτήτε που δραστηριοποιούνται σε αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνες είναι διαθέσιμα για τις εθνικές αρχές για του στόχου εφαρμογή. Τη συμφωνία όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και δεν μπορούν να δημοσιευθούν. Για όλους τους υπόλοιπου σκοπούς είναι δυνατή η χρήση τους. Σα ευχαριστούμε μάλιστα κυρία Λεβίν. Ε, όμως αρχίζει έτσι το άρθρο. Τα μέρη θα μεριμνήσουν ότι ε, ώστε η αδίποτε στιγμή όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με ευρωπαϊκά σκάφη και τι αλληλευτικέ δραστηριότητε στα ύδατα του Μαυρικίου θα θεωρούνται διαβαθμισμένα. Μπορείτε να τη διαβάσετε αυτή την πρόταση. Οτιδήποτε σχετίζεται με τα σκάφη και τι δραστηριότητε, όλα είναι εμπιστευτικά τα στοιχεία. Και στην επόμενη πρόταση από αυτή που διαβάσατε εσεί είναι η ίδια όπω τελειώνει και το άρθρο. Δηλαδή, Κατά τη γνώμη μου, όπως δερμηνεύω εγώ τη διατύπωση, τίποτα δεν θα αποκαλυφθεί σε κανένα τρίτο μέρος που επιθυμεί να γνωρίζει τα περί αλλιευτικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένες και της κοινωνίας των πολιτών του Μαυρικίου. Αυτό είναι ένα πράγμα δεύτερο οι πληρωμές που λαμβάνουν οι πλειοκτήτες. Ε, μα μιλάμε για το ίδιο ακριβώς ποσό που βλέπουμε από πότε, ούτε καν θυμάμαι, 2002, κάτι τέτοιο, 35 ευρώ ο τόνος. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Ε, εγώ νόμιζα ότι με τη νέα συμφωνία μιλούσατε για συμφωνίες νέας γενιάς ε, και ήλπιζα ότι θα αυξάναμε τις αμοιβέ των πλειοκτητών. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί δεν έγινε αυτό. Ευχαριστούμε ο κύριος Σάντσες. Ε, Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ή δύο σχόλια δεδομένων των παρατηρήσεων της κυρίας Λέβεν. Δεν ξέρω κατά πόσο με κατάλαβε σωστά, παρότι προσπάθησα να είμαι σαφής. Είπα σαφώ ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατηγικό έγγραφο, χωρών και σε αυτό το έγγραφο λέει ότι η δημοκρατία της Μαυριτανίας συμπεριφέρεται καλά όσον αφορά το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει συχνά στις διαβουλεύσεις όταν μιλάμε για πολιτικές και ούτω καθεξής. Και ότι η ο κόσμος συμμετέχει σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος. Αυτό αναγράφεται μέσα στο έγγραφο της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω λάβει διαμαρτυρίες από οργανισμούς ε, από τη δημοκρατία της Μαυριτανία όσον αφορά το επίπεδο διαφάνειας. Γι' αυτό το λόγο το θέτω αυτό στην Κομισιόν, διότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διαφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για το Μαυρίκαιο όπως και για τη Μαυρίτανία υπάρχουν ε, ιδιωτικέ ε, συμφωνίες και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές οι συμφωνίες. Πρέπει να δούμε τις μελέτες αντικτύπου φαίνονται πολύ λεπτομερείς και αναλυτικές και εξετάζουν πολλά και διάφορα ζητήματα. Μία πτυχή αφορά την εμπιστευτικότητα, διαβάθμιση. Όταν μιλάμε λοιπόν για εμπιστευτικότητα και διαφάνεια. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία της εμπιστευτικότητας που δεν επηρεάζουν τη διαφάνεια. Για παράδειγμα σε βιομηχανικές δραστηριότητες, η βιομηχανική τεχνογνωσία, τεχνικές γνώσεις, μια βιομηχανία νόμιμα μπορεί να προστατεύει κάτι τέτοιο εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την υλοποίηση, την εφαρμογή της συμφωνίας και ορισμένες ε, διατάξεις. Αν υπάρχει συγκεκριμένη τεχνογνωσία ε, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται, αλλά ορισμένα άλλα πράγματα είναι δύσκολο να τα κανεί σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Και εγώ είμαι υπέρ τη διαφάνεια. Πολύ γνώση μπορεί να δημοσιοποιηθεί και πρακτική με τρόπο μη επίσημο, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό γίνεται με κάποια ισορροπία. Όσον αφορά την περιφερειακή προσέγγιση, πάντα έλεγα ότι είμαι υπέρ, αλλά από το 2007 και μετά υπήρχε μια συμφωνία, ε, δεν υπήρχε μια συμφωνία, συγγνώμη, και ξαφνικά περνάμε σε μια προσέγγιση η οποία είναι επιθυμητή αλλά ίσως όχι ρεαλιστική αυτή η περιφερειακή προσέγγιση. Για να έχουμε μια περιφερειακή προσέγγιση πρέπει να έχουμε μια ικανοποιητική συμφωνία και ένα ικανοποιητικό πρωτόκολλο. Και μετά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον όσον αφορά τις τιμές πιστεύω έχουν ε, βελτιωθεί ευνοϊκά οι όροι σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο. Φυσικά υπάρχει, υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους όρους και τις συνθήκες και ειλικρινά ε, είναι εξωφρενικό εφόσον οι αντισυμβαλόμενοι είναι ικανοποιημένοι με αυτές τις πτυχές γιατί εμείς να προσπαθούμε να ζητάμε περισσότερα ώστε να επιτύχουμε τα ίδια. Εμείς πάντα δρούσαμε σωστά με τον Μαυρίκιο και τα οικονομικά επίπεδα ήταν πάντα πολύ ψηλά. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια, αν όχι, ας περάσουμε. Στο επόμενο, ο εκπρόσωπος της θέλει το λόγο. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα των συμφωνιών ε, νέας ε, γενιάς. Ε, πρέπει να θυμόμαστε από τι αποτελείται από 4-5 διαφορετικά τμήματα αυτή η συμφωνία. Καλύτερη, καλύτερα επιστημονικά στοιχεία. Αυτό το καλύπτουμε. Να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία το, του Διεθνού Ινστιτούτου για τον τόνο ή για τα στοιχεία της Οικονομικής και Τεχνικής Επιτροπής. Το κάναμε αυτό. Μιλάει για κλαδική στήριξη. Το κάναμε αυτό. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κάναμε και αυτό. Η φιλοδοξία μας είναι να αυξήσουμε με ε, την συνεισφορά προς την βιομηχανία μέσα σε αυτές ε, τις ε, συμφωνίες. Δεν γίνεται όμως αυτό νυχθημερών και για την περιφερειακή προσέγγιση αυτό είναι τμήμα της περιφερειακής προσέγγισης. Πρόκειται για άκρος μεταναστευτικά είδη και άρα εγγράφεται πλήρως στο πλαίσιο και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί βάσει της συμφωνίας δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το θέμα της πρόσβασης. Υπάρχει και η κλαδική συνιστόσα που είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσα στη συμφωνία και θα πρέπει να είναι υποφελές για ε, ε, ολόκληρο τον κλάδο, όλους τους φορείς ε, του κλάδου, όχι ένα συγκεκριμένο τμήμα του στόλου. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα περάσουμε στο σημείο 11 ε, συμφωνία αλλιευτική σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης ε, και στις 19 Νοεμβρίου μας παρουσίασε το νέο πρωτόκολλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ριβελίν που είναι ο εισηγητής μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία Αλλιευτικής Σύμπραξη που συνήθει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Μαδαγασκάρη επιτρέπει σε ευρωπαϊκά αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν στα ύδατα της Μαδαγασκάρης και ενταστεί στη σειρά αλλιευτικών συμφωνιών που συνάπτονται με τις χώρες του Ινδικού ωκεανού. Το πρωτόκολλο το οποίο δημιουργεί τη δυνατότητα αλλιευσής από ευρωπαϊκά σκάφη και ορίζει το χρηματικό αντίτιμο λίγη το Δεκέμβριο του 2012. για αυτό το λόγο χρειάζεται ένα νέο πρωτόκολλο κατάλληλο για τις δυνατότητες και τις απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Στόλου. Θα πρέπει να συναφθεί ένα τέτοιο πρωτόκολλο το συντομότερο. Εγώ προτείνω η Επιτροπή Αλίας να δώσει την έγκρισή της για σύναψη νέα ε, συμφωνίας αλληλευτικής σύμπραξης για περίοδο 2 ετών 2013-2014 και που να προβλέπει δυνατότητες αλλιευτικές για 96 σκάφη 54 θυναλιευτικά και 56 ε, παραγαδιάρικα με χρηματικό, χρηματική αντιπαροχή πλήρη. Ίση με 3.050.000 ευρώ με αύξηση 328.000 ευρώ το χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία από το 2007 μέχρι το 2012. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει 975.000 ευρώ για πρόσβαση στην αλληλευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης που αντιστοιχεί σε ε, ποσότητα ε, αναφοράς 15.000 τόνων το χρόνο. Μιλάμε για 1.700 τόνους περισσότερους σε σχέση με την προηγούμενη και 550.000 ευρώ το χρόνο για την πολιτική ανάπτυξη της Ελίας στη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης. Η αύξηση των ποσών σχετίζονται με μια αύξηση χρηματικού ε, χρηματικής αντιπαροχής εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η αύξηση των αλλιευμάτων συμμορφώνεται πλήρως με τις καλύτερες επιστημονικέ γνωμοδοτήσει τη επιτροπή Τόνου του Ινδικού ωκεανού. Ωστόσο, όσον αφορά τη χρήση στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας Ελευτικής Σύμπραξης, τη χρήση των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην Ευρώπη, στην εταιρεία Μαλγκάς, για την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια, που χρηματοδοτεί την εθνική πολιτική αλληλείας, είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι οικονομικοί εξωτερικοί έλεγχοι, audit δηλαδή, ώστε να υπαλληθεύονται οι δηλωθήσεις δαπάνες. Τέλος, όσον αφορά την πολιτική κατάσταση στη Μαδαγασκάρη, παρά κάποιες εντάσεις ε, απομένει γεγονός ότι η διαδικασία για να τεθεί τέλος στην κρίση της Μαδαγασκάρης όπως υπογράφηκε το 2011 τηρείται και παραμένει το πλαίσιο αναφοράς για την αξιολόγηση των ιστορικών ε, εξελίξεων στη χώρα. Οι επόμενες εκλογές θα λάβουν χώρα τον ε, Μαΐο και Ιούλιο του 2013 παρουσία παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια εκλογική επιτροπή ανεξάρτητη έχει ήδη οριστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος θα ήθελε να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει. Δίνουμε το λόγο πρώτα στην Επιτροπή, όπως κάνουμε συνήθως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που είναι υπέρ τη συμφωνία αυτή. Ο κύριο Συγητή είναι σημαντική. Επίση, αποτελεί το αντικείμενο διαπραγμάτευση σε πολύ δύσκολο πλαίσιο. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση, την κατάσταση στη Μαδαγασκάρη. Πρόκειται για μια συμφωνία που διαπραγματευτήκαμε σε στενή συνεργασία με του συναδελφού μα στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, τόσο ω Βρυξέλλε όσο και εκεί επιτόπου και φυσικά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε σχέση με το άρθρο 96 της διαδικασίας Κοτονού και όλα αυτά αντιπροσωπεύονται όπως και η προηγούμενη συμφωνία ε, περιλαμβάνει τι βασικέ αρχέ μεταρρυθμίσει. Έχουμε τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε το διαχωρισμό τομέακων στηρίξεων από το τέλο πρόσβαση. Έχουμε την αιρεσιμότητα σε σχέση με αυτό. Και φυσικά συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή του Ινδικού Ωκεανού και την Επιστημονική Αρχή την Επιστημονική Επιτροπή τη, ώστε να βασίσουμε τι ποσότητέ μα στι δικέ του συμβουλέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπεσέρ. Ναι, ευχαριστώ. Ε, έχω κάποιους ενδιασμούς για αυτό το πρωτόκολλο, για το περιεχόμενό του, όχι για την ανάλυση του που με κάνει να το θεωρώ αρκετά θετικό, αλλά με ανησυχεί το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται όπου υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες όσον αφορά την εφαρμογή του. Λοιπόν, αυτό το πρωτόκολλο κατά την άποψή μας είναι μάλλον άριστο. Άρτιο συμμορφώνεται μάλιστα χρονικά με την εκθέση που εγκρίναμε πριν λίγες μέρες ε, στο Στρασβούργο με τη φίλη και συνάδελφο Ιζαμπέλα για την εξωτερική πολιτική της αλληλευτικής πολιτικής. Οι αρχές ε, μας ικανοποιούν, οι συστάσεις ε, ε, η αλληλεία βασισμένη σε συστάσεις επιστημονικές που υπάρχουν διαθέσιμες μια, ένα κομμάτι του αντιτίμου που θα υποστηρίζει την παραδοσιακή αλληλεία, την τομεακή αλληλεία της Μαδαγασκάρης ευρωπαϊκή στόλη που δεν θα είναι ανταγωνιστική με τον εθνικό στόλο της Μαδαγασκάρης ενίσχυση των ελέγχων της παράνομης αλίας, ε, πολύ ενδιαφέρον και ε, νέα μέτρα για την προστασία των καρχαριών σε αυτό το χώρο. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα μικρό πρόβλημα και πάλι το θέμα της εμπιστευτικότητας την οποία ξαναβλέπουμε εδώ όπως συζητήθηκε προηγουμένως ε, για την δημοκρατία του Μαυρικίου και αυτή η συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη περιλαμβάνει μια ρήτρα εμπιστευτικότητα. ίδια φύση με εκείνη που έχουμε για το Μαυρίκιο. Μάλλον καλά είναι όλα αυτά. Προφανώ, όπω είπε και ο συζητητή, θα έπρεπε να μα οδηγήσουν όλα αυτά να είμαστε υπέρ, ιδιαίτερα ευνοϊκοί προ αυτό το πρωτόκολλο, αλλά έχουμε ένα πολιτικό χρονοδιάγραμμα, αδιαμφισβήτητο με τις εκλογές. Έχουμε μια εγγύηση που θα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στείλει παρατηρητές κατά τη διάρκεια αυτών των εκλογών. Αλλά γνωρίζουμε πόσο εύθραστη είναι η δημοκρατία στη νήσο Μαδαγασκάρη. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Η αιρεσιμότητα αυτή για τη δημοκρατία διασφαλίζεται. Τι διασφάλιση έχουμε εν τέλει ότι αυτή η συμφωνία όσο καλή και αν είναι μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί λόγω υποβάθμισης της πολιτικής κατάστασης στη Μαδαγασκάρη. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην Ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, αλλά πρώτα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να κάνω μια ερώτηση. Σύμφωνα με πληροφορίε που έχω λάβει εγώ, έγινε μια αλλαγή στην νομική βάση όπω φαίνεται Αντικαθιστούμε το 43-2 με το 43. Ε, μια ερώτηση είναι αναπάντητη ως προς το τι θα κάνει η Κομισιόν. Θα μπορούσατε να μας το απαντήσετε τώρα. Επίσης, ποια θα είναι η τοποθέτηση της Κομισιόν όσον αφορά τη νομική βάση αυτής της ε, συμφωνίας και του πρωτοκόλλου. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να επανέλθω στο θέμα των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, για μας ε, όντως δεν υπάρχουν εχέγγυα. Είναι ξεκάθαρο αυτό στην ε, μεταβατική φάση. Έχουμε το, άρθρο, το νοδικό χάρη του άρθρου 96. Επίσης συνεργαζόμαστε με την Μαδαγασκάρη για να ακολουθήσει την δημοκρατική οδό ε, και θέλουμε να παραμείνει σε αυτό το δρόμο στον οποίο επέστρεψε και το πρώτο εξάμεινο του 2013 θα γίνουν εκλογές. Έχουμε δέσμευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής ένωση να χρηματοδοτήσει εν μέρη την εκλογική αυτή αναμέτρηση. Θα αποστείλει και παρατηρητές η Ένωση. Τρόπον την η κατάσταση που επικρατεί εκεί δεν διαφέρει από την κατάσταση που διαπιστώνουμε σε άλλες χώρες με ευαίσθητα ε, δημοκρατικά διαπιστευτήρια. Ε, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν ήσασταν εδώ καν, το 1998 έγινε πραξικόπημα στη Μαυριτανία, παραδείγματος χάρη, ε, και τότε δεν είχαμε καμία ρήτρα για ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε και είχαμε μέσα στη διάθεσή μας για να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε ε, πίεση, ούτως ώστε να εξέλθουν από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αντίθετα, έχουμε δύο τέτοιες ρήτρε ε, αναβολή και αναθεώρηση των οικονομικών εισφορών, άρθρο 8 γάμα, ιδιαίτερος που, λέει, που μας δίνει τη νομικό στη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό όταν έχει σημειωθεί παραβίαση των βασικών ε, ε, δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει και τη Συμφωνία Κοτονού. Ε, και στη συνέχεια έχουμε τη ρήτρα αναστολής της εφαρμογής ε, της ίδιας συμφωνίας. Ε, δηλαδή αν καταγγείλει την συμφωνία ένα από τα μέρη για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 9 της Συμφωνίας Κοτονού πάλι προβλέπεται διαδικασία. Δηλαδή τώρα είμαστε εξοπλισμένοι σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να δώσουμε άλλε εγγύσει, αλλά πάντως αυτό αποδεικνύει ότι είναι σοβαρό το ζήτημα για μας. Ας επανέλθω τώρα στο θέμα της νομικής βάση ε, ε, Έχουμε τρία ε, ε, στοιχεία στο παζλ σε σχέση με όλες αυτές τις συμφωνίες και σύμπραξη, οικονομικές συμφωνίες και τα λοιπά. Σε σχέση με την φύση των νομοθετημάτων, ε, λοιπόν, έχουμε διαφορετικές διαθέσιμες νομικές βάσεις. Ένα είδος απαιτεί την συγκατάθεση ε, προποθέτει μάλλον την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ώστε να χρησιμοποιείται η κατάλληλη νομική βάση και με επιστολή του ίδιου του Επιτρόπου που κοινοποιήσαμε ε, στην Επιτροπή προβλέπεται ότι για τη σύναψη πρωτοκόλλου ή για συμφωνία ελευθέρου εμπορία χρησιμοποιείται το ε, Άρθρο 43.2 και το 183.6 εδάφιο 2 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης. Ε, η, Επιτροπή ανέκαθεν ήταν ερήτη και κατηγορηματική για αυτό το θέμα σε οποιαδήποτε συζήτηση έγινε σε οποιοδήποτε βήμα. Αν ε, χρησιμοποιηθεί ακατάλληλη νομική βάση για οποιοδήποτε νομοθέτημα τότε όταν και αν συμβεί αυτό, αλλά να έχει συμβεί, ε, θα αναθεωρεί στην κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή πρέπει να έχει συνάψει τη συμφωνία το Συμβούλιο. Πάντως ο θεσμικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβώς να μεριμνώσει να χρησιμοποιεί την κατάλληλη νομική βάση. Είμαστε και θεματοφύλακε τη συνθήκη, μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά πάντω εμεί είμαστε μετακίνητοι και ξεκάθαροι για τη θέση μα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε ή όχι δεν έχω να προσθέσω τίποτα, δεδομένου ότι συμφωνούμε με τον συνάδελφο όσον αφορά την τεχνική καλατιλότητα της συμφωνίας. Τώρα όσον αφορά το πολιτικό ζήτημα της Μαδαγασκάρης, το πίνακα του Μαρτίου που υπάρχει εδώ και που μου την έστειλαν ε, τήρηται μέχρι στιγμής. Πιστεύω λοιπόν ότι η γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι ευνοϊκή. Φυσικά καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τους εξωτερικούς οικονομικούς ελέγχους ώστε οι δελωθείς δαπάνες να κατευθύνονται πράγματι προς τους στόχους να δρομολογούνται προς τους προτινόμενους στόχους. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριβελίνη. να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο τη της διάταξη, σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχουμε μία γνωμοδότηση με εισηγητή τον κύριο ε, Ριβελίνη και η Επιτροπή είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε, μιλάμε για Ανταρκτική, Καραϊβική, Ατλαντικό και Ινδικό ωκεανό και Ειρηνικό ωκεανό. Και αυτά τα εδάφη εξαρτώνται συνταγματικά από τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Δανία, Γαλλία, Κατοχώρες και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αναθεωρήσει τις αρχές που εμπνέουν τη συνεργασία της με αυτές τις χώρες. Αυτή η νέα προσέγγιση θα πρέπει να ευνοήσει την αεφορονάπτυξή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιοχών του Ατλαντικού, της Ανταρκτικής, της Καραϊβικής, του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού θα πρέπει να συμβιβάζει τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες όπως δατοκολίεργεια και αλληλεία, τουρισμό, ε, ναυτιλία ε, με τη χρήση ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, λαμβάνοντα υπόψη τις ε, ανθρώπινες δραστηριότητες και τα ε, θέματα του κλίματος. Σε θέματα αναυσιπλοείας, η συνεργασία θα πρέπει να προωθεί τη γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοτεχνολογίας, της ωκεάνιας ενέργειας, της θαλάσσιας επιτήρηση, τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και τη διαχείριση βάση οικοσυστημάτων όσον αφορά την αηφόρο διαχείριση των η αποθεμάτων, η συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε υπεύθυνη διαχείριση της αλληλείας στο πλαίσιο της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των ηχθή αποθεμάτων με τακτική διαβούλευση μεταξύ των δύο μέρων όσον αφορά τη διατήρηση, τη διαχείριση των βιολογικών και θαλάσσιων πόρων και με ανταλλαγές πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση των πόρων. Όσον αφορά το τομέα της η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρέπει σε μεγάλο βαθμό να υποστηρίξει τα τοπικά συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης, ώστε να καταπολεμήσει την παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλληλεία και το σχετικό εμπόριο. Επίσης είναι αναγκαία αποτελεσματική συνεργασία με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης τη αλληλείας και με αυτές ώστε να καταπολεμηθεί η λαθρέα και παράνομη αλληλεία που σήμερα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές της βιωσιμότητας των αλληλευτικών αποθεμάτων, πόρων και της βιωσιμότητας των ωκεανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να ενισχυθεί ο συντονισμός και η συνεργασία, για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παράνομη αλληλεία, εγώ σκοπεύω να υποβάλω μια τροπολογία που θα τροποποιεί το άρθρο 19.2β της πρότασης της ε, Κομισιόν και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω ακριβώς λεπτομέρειες και να σας το διαβάσω και να σας το τεκμηριώσω επίσης. Ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη. Δύο εκπρόσωποι είναι εδώ από την ε, Κομισιόν, ο κύριος Σαλαμάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορέσαμε να δεχτούμε την πρόσκληση της Επιτροπής σα για να σας παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν για μια απόφαση σύνδεση των υπεράκτων εδαφών ε, των εξόχως υπερπόντιων χωρών και εδαφών και αποτέλεσαν αντικείμενο ζητήσεων στο Συμβουλίο. Ο εισηγητής σας, ο κ. Ριβελίνη, πολύ σωστά παρουσίασε τις πτυχές που αφιερώνει αυτή η πρόταση απόφασης στα ζητήματα που σχετίζονται με την αλληλεία, με τις αλληλευτικές δραστηριότητες, αλλά και όσον αφορά τις παρακτές περιοχές. Θα ήθελα, αν μου το επιτρέπετε, με λίγα λόγια να υπενθυμίσω το πλαίσιο στο οποίο εντάξεται αυτή η πρόταση απόφασης και στο οποίο την μελετήσαμε. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε μία απόφαση ε, συνεργασίας του 2001. Υπήρχε λοιπόν λόγος να αναθεωρηθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές, οι μεταβολές που έχουν λάβει η χώρα από τότε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπερπόδιες χώρες και τα εδάφη Ξεκίνησα μια περίοδο προβληματισμού που ξεκίνησε το 2008 μια πράσινη βίβλο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολούθησε δημοσία διαβούλευση ενός έτους η οποία έδωσε συνέχεια σε μια ανακοίνωση το 2009 Στη συνέχεια στο 2010, το Δεκέμβριο, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα για τις προτάσεις της Κομισιόν στην ανακοινωσή και κάλεσε την Κομισιόν να παρουσιάσει μια νέα πρόταση απόφασης το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Οι 26 υπερπόντιες χώρες και τα τέσσερα κράτη-μέλη που σχετίζονται με αυτές υπέβαλαν μια κοινή τοποθέτηση το Μάρτιο του 2011 στην οποία συνόψησαν τις φιλοδοξίες τους σε σχέση με την εξέλιξη αυτή τη συνεργασία τη Ένωση, τη σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερπονίων χωρών και εδαφών. Σε αυτό το διάστημα είχαμε επίση την ευκαιρία ανταλλαγή με όλους τους ενδιαφερομένους σε διάφορα φόρουμ και σε πλαίσια πολιτικού διαλόγου όπω προβλέπονται από την απόφαση σύνδεση, αλλά και στη διάρκεια πολλών τεχνικών συνεδριάσεων, τριμερών με τους εκπροσώπους αυτών των εδαφών και εκπροσώπους των τεσσάρων κρατών μελών. Η πρόταση που διαβιβάσαμε θεωρούμε ότι είναι ταυτόχρονα φιλόδοξη και ρεαλιστική. Οι στόχοι που προσδιορίζει περιλαμβάνουν την καθιέρωση στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ ε, των υπερπόντων χωρών και εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολό τους, μέσω μεταξύ άλλων της ανάπτυξης εμπορικών δικτύων. Ένα θέμα που θα σας αναπτύξει ο κ. Βάλς σε λίγο. Άλλος στόχος, η καθιέρωση πιο αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε βασισμένων σε κοινέ αξίες η βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα των υπερπόντων χωρών και εδαφών. Τέταρτο στόχο, ενίσχυση τη ε, δυνατότητα του προσαρμογή και η μείωση τη ε, βάλω του χαρακτήρα του ε, συνεργασία των υπερπόντων χωρών και εδαφών με τρίτους εταίρους τους και τέλος η πρόθεση αξιών, προτύπων και συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Αυτή η πρόταση απόφασης προσφέρει, αποτελεί ουσιαστικά τη νομική βάση, την απαραίτητη νομική βάση για δράσεις σε τομείς που οριστήκαν ως τομείς προτεραιότητας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η έννοια του αμοιβαίου συμφέροντος μπορεί μερικές φορές να προκαλεί σύγχυση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτός ο όρος δεν σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε από τις ανάγκες των υπερποντών χωρών και εδαφών σε θέματα ανάπτυξης. Αυτή είναι, κατά την άποψή μας, καθιερώνει μάλλον έναν σταθερό σύνδεσμο με τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες των υπερποντων χωρών και εδαφών. Δεν θα επιτρέψει ωστόσο παράληψη άλλων τομέων. Μίλησα για την αποφάση του 2001, η οποία εκείνη την εποχή είχε σκοπό τον εξυγχρονισμό. Συμπεριλάβουμε κάποιες, ε, όπως θεωρούμε, βασικές καινοτομίες. Πρώτον, θελήσαμε να αφιερώσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι στον τομέα της συνεργασίας. Με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών. Αυτό το μέρος περιλαμβάνει επίσης τα άρθρα που αφορούν την αλληλεία, τους αλληλευτικούς σπόρους και τις παράκτιες περιοχές. Το άλλο κομμάτι της πρώτης απόφασης σχετίζεται με το εμπόριο και τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το εμπόριο. Εκεί προτείνουμε μια σειρά νομικών διατάξεων που συνεχίζουν να προσφέρουν ένα εμπορικό καθεστώς ε, ιδιαίτερα προνομιακό προ όφελο των υπερποντών χωρών και εδαφών και που ανταποκρίνεται στι ανάγκε βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, Τέλο, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην περιφερειακή συνεργασία. Εμεί προτείνουμε σημαντική αύξηση του περιφερειακών κονδυλίων σε σχέση με το τι γινόταν στα προηγούμενα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά ταμεία. Αυτό που δεν αλλάζουμε και το οποίο διατηρούμε είναι η αρχή της προγραμματι... προγραμματίσιμης βοήθειας καθώς και τον κανόνα για τον τομέα συγκέντρωσης ώστε να είναι αποτελεσματική η χρηματοδοτική αρρωγή της Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, εν συντομία, αυτό είναι το περίγραμμα αυτής της πρώτης απόφασης δώσω το μικρόφωνο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση αυτή συνοδεύτηκε από ανάλυση αντικτύπου ιδιαίτερα λεπτομέρη που ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να διαβάσουν τα... Ε, οι εδώ και σε κάθε είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής και του κ. Ζηγητή, του κ. Ριβελίνη για να σας παρέχουμε οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριος Δράνκοβελ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το εμπορικό καθεστώς που θεσπίζει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου, η απόφαση και για την απόφαση που λάβαμε τι θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει εσάς εδώ στην Επιτροπή Αλίας. Τρεις είναι οι καινοτομίες. Πρώτον, ενισχυμένες, ε, ενισχυμένοι όροι και κανόνες προέλευσης για τις εξαγωγές προς υπερπόδια εδάφη, απρόσβαση στις υπηρεσίες και τρίτον, εστίαση στα εμπορικά ζητήματα και αν μου το επιτρέπετε θα ήθελα να ε, επικεντρωθώ στο πρώτο σημείο. Από το 1991 η απόφαση του Συμβουλίου αυτή χορήγησε φορολογική ατέλεια και απουσία δασμολογικών ποσοστώσεων για τα υπερπόντια εδάφη και χώρες. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, απλώς ε, προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους για να βελτιώσουμε το καθεστώς και βρήκαμε τρεις τρόπους για να το κάνουμε αυτό. Πρώτον, εξυγχρονισμός και ενίσχυση των κανόνων ε, προέλευσης. Δεύτερον, ε, διευκρίνηση των κανόνων τους ώστε να είναι εύρυθμη πρόσβαση στην αγορά για διοικητικούς λόγους, ε, για τις παρατυπίες, ισχύουν οι τυπικές διαδικασίες που γνωρίζετε πολύ καλά. Δεύτερον, ζητήθηκε η απουσία διακριτικής μεταχείρισης σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές ε, Βραζιλία, Ινδία και Κίνα συγκεκριμένα. Για τους κανόνες ε, προέλευσης ε, και γνωρίζω πόσο σας ενδιαφέρουν, θα ήθελα να προσθέσω κάποιες λεπτομέρειες. Στην διαβούλευση εντοπίστηκε αυτή η θεματική ενότητα ως ένας τομέας όπου επιδέχονται βελτιώσει κανόνες προέλευσης που ως επιτοπλίστων χρονολογούνται εδώ και 11 12 χρόνια, οπότε προτείνουμε ένα νέο σύστημα ε, κανόνων προέλευσης για το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων, το GSP. Απλουστεύουμε με τους νέους ε, κανόνες ε, ή απαλύνουμε τους κανόνες κυρίως για τα ελευτικά προϊόντα και θα ήθελα να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να διαπιστωθεί η προέλευση του ψαριού, παραδείγματος χάρη, ή μάλλον η σημαία του αλευτικού σκάφους δεν θα χρειάζεται πλέον ε, το πλήρωμα να πληρεί συγκεκριμένε απαιτήσει ε, περί εθνικότητας, δηλαδή να είναι υπήκοοι των ε, υπερποντίων χωρών και εδαφών. Αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς βάσει του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων. Δεύτερον, οι νέοι κανόνες για την επιστοποίηση της προέλευσης των καταγεγραμμένων εξαγωγέων. Η αυτοπιστοποίηση επωνομαζόμενη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βελτίωσης που προτείνουμε. Τις λεπτομέρειες θα τις έχετε αν θέλετε μέσα στο έγγραφο, αλλά είμαι και εδώ στη διάθεσή σας αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελε κάποιος το λόγο. Κύριε Πυρελίνη, όχι. Ωραία. Θα σε ευχαριστούμε τότε και πάμε ε, στο ε, επόμενο σημείο, δηλαδή εκθέσεις σχετικά με την αντιπροσωπεία τη επιτροπή Αλίας στη Βενετία 9 με 11 Οκτωβρίου 2012. Έχετε από τη γραμματεία το σχετικό σημείωμα. Ο κύριος Στίβενσον που ήθελε το λόγο δεν είναι εδώ και ούτε ο πρόεδρος ε, της αποστόλης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος για να μας μιλήσει για αυτό το σημείο. Έχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, όχι λοιπόν. Οι δύο αρμόδιοι λείπουν, οπότε θα περάσουμε, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις στο επόμενο σημείο, δεν υπάρχουν, πάμε στο 14, έκθεση σχετικά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αλίας ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλίας ε, στο Βίγκο, Ισπανία. Και γι' αυτό το θέμα έχετε μία περίληψη στους ε, φακέλους σας. Sí, señora García Ούτε εδώ είναι ε, παρόντες ε, οι αρμόδιοι. Παρακαλώ, κυρία Γκαρσία Ερέιρο. Μετά ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής που μας βοήθησε στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Αλλά πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά θετική. Αυτό το διήμερο ήταν με ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα. μισή ημερών δουλειά κάναμε σε δυόμιση μέρες ουσιαστικά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι καταφέραμε να αντιληφθούμε ότι όσοι εργάζονται σε αυτά τα λειτουργικά προγράμματα, στον έλεγχο και την επιθεώρηση μαζί με τα κράτη-μέλη, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των οργανισμών, του οργανισμού. Πιστεύω ότι γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Συζήτησαν μαζί μου, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επειδή ορισμένες φορές δεν έχουν αρκετά στοιχεία ώστε να μπορούν να προχωρήσουν, να σημειώσουν πρόοδο σε ορισμένου τομεί, ειδικότερα τους τομείς που σχετίζονται με το ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας πολιτικής. Και εδώ για να αναφέρω απλά τη δέσμευση που έγινε. Ο οργανισμός έχει 57 άτομα προσωπικό. Υπάρχει κατάρτιση, ο έλεγχος, οι πτυχές θαλάσσιου ελέγχου και έχουν ένα προπολογισμό, ένα κονδύλιο προπολογισμού που δεν τους επιτρέπει να υλοποιούν όλες τις πτυχές ελέγχου. Το κονδυλίο για αυτή την πτυχή έχει αφαιρεθεί και μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό για τα κράτη-μέρη να υπάρχουν κονδύλια διαθέσιμα γι' αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τα πάντα υπό τις δύσκολες σημερινές περιστάσεις αλλά μου φαίνεται ότι πιστεύω εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο του οργανισμού αυτού. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο κατάρτιση. για να εκπαιδεύουν επιθεωρητές. χρειάζονται περισσότερα. ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και πιστεύω το ολοκληρωμένο σύστημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο να μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια και αυτό πιστεύω ότι είναι κρίμα Είναι κρίμα που είμαστε τόσο λίγοι εδώ, γιατί το ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό. Είναι σημαντικό όλοι μας να καταλάβουμε καλύτερα το έργο συνεργασίας και ανάπτυξης που λαμβάνει η χώρα εδώ. Πραγματικά συμφωνεί τα όσα παρουσιάζουμε εδώ σε αυτήν την Επιτροπή. Ο κύριος Ντέβις, παραδέχομαι ότι όταν πήγα στο Βίγκο ήμουν λίγο κοινικό σε σχέση με το έργο αυτή, αυτού του οργανισμού ε, και σταδιακά άλλαξα γνώμη. Μίλησα με τους επιθεωρητές, ε, στελεχώνεται ο οργανισμός από επαγγελματικά επαρκείς ανθρώπους ε, που δουλεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξέρουν τα πάντα, τα, όλα τα κόλπα των ψαράδων τα ξέρουν. Και και η εντύπωση που μου έδωσαν είναι ότι όλο ένα και περισσότερο αναδεικνύονται σε ένα πυρήνα δικτύου ανταλλαγής βελτίστων ε, πρακτικών και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που, έχουν, ε, που υπάρχουν για να, την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Good information now, τα ημερολόγια του πλοίου, τα ε, στοιχεία από τους δορυφόρους, ε, ε, είναι δυνατή παρακολούθηση αλλιευτικών σκαφών σε πραγματικό χρόνο μέχρι τελευτα... δηλαδή κάθε λεπτό και μπορούμε να δούμε και την πρόοδο στη συνέχεια για να ξέρουμε ε, τι συμβαίνει ακριβώς και οι επιθεωρητές ε, που ε, κάνουν καλά τη δουλειά τους μπορούν να ταυτοποιήσουν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση. Άμα εξαφανιστεί για μία ώρα το σκάφος, αυτό συμβαίνει με τον κινέζικο στόλο, ένα μίλι παρακάτω, ε, μπορεί να γεννηθούν κάποια ερωτηματικά σε σχέση με τα αλληλευόμενα αποθέματα. Όχι, εντυπωσιάστηκα πρέπει να το πω και ε, ο οργανισμός ελπίζω να συνεχίσει να αναπτύσσει αυτό το ε, κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε όλους τους επιθεωρητές όλης της Ένωσης δηλαδή και δεύτερον λένε και περισσότερο αποκτά πρόσβαση ε, σε δεδομένα από άλλες ευρωπαϊκές πηγές χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει για αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία στο έπακρο, πρέπει να προσέχουμε και τον προπολογισμό, μην το ξεχνάμε. Ε, διότι πρόκειται για κοινό πόρο όλων των κρατών ε, που έχουν ε, αλλιευτικούς σκόφους. Γίνεται χρηστή χρήση των κονδυλίων. Δηλαδή κάτι να πω μόνο για τους επιθεωρητές. Όταν μπορούν όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάτι έκνομο, μια παρατυπία, κάτι που δεν συνέβη με το βασικό κανονισμό, ε, ε, κάνουν την καταγγελία σε ένα φάκελο, φροντίζουν ώστε να δοθεί μια συνέχεια και να ακολουθήσει η δίωξη από τις αρμόδιες αρχές. Ωραία όλα αυτά. Μετά τι γίνεται, προβλέπει η νομοθεσία ότι για το ποινικό δίκαιο ε, είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη και πρέπει να είναι αποτρεπτικά και ανάλογα τα μέτρα. Αλλά αυτό πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και αν είναι τώρα να έχουμε χρονοβόρα και έρευνα με σκάφη περιπολίας ε, και το αποτέλεσμα είναι ε, να χτυπήσουμε, να, να τιμωρήσουμε με ένα χαστούκάκι το, ε, το κράτος μέλος που έχει παρατυπήσει δεν νομίζω ότι ωφελεί. Δηλαδή θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο ε, εφαρμόζω, την νομοθεσία από τα κράτη-μέλη. Ε, δεν μιλώ για επιβολή ε, ομοιόμορφων ποινικών κυρώσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τουλάχιστον να φροντίσει η Επιτροπή να είναι τα επίπεδα, μάλλον να εισηγηθεί ποια θα ήταν τα καταλληλότερα, ποιε θα ήταν οι καταλληλότερε κυρώσεις. Ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντσες ως ε, μέλος της αντιπροσωπείας ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Συμφωνώ πλήρω με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι ότι πρόκειται για ένα πολύ θετικό και ενδιαφέρον ταξίδι. Κατά την άποψή μου τρει ήταν πτυχέ που είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η πρώτη είναι τα κοινά σχέδια που καταρτίζονται για τα διάφορα είδη και για τις αλλαγές στον οργανισμό στο μέλλον αυτά τα σχέδια θα πρέπει να έχουν μια πιο περιφερειακή διάσταση. Υπάρχουν ήδη σε διάφορα ύδατα και η πραγματοποίηση ελέγχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μπορούμε να χρησιμοποιηθούν μάλλον ε, αυτά για τον έλεγχο τη αλληλεία των ελευθερικών δραστηριοτήτων, ώστε να παρέχουν περισσότερε πληροφορίε. Το δεύτερο είναι ότι θα μπορούσε να αποτελεί το κέντρο και κομβικό σημείο για τη λήψη δεδομένων, στοιχείων, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τι αλληλευτικέ δραστηριότητε και την αλληλεία. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τη διαχείριση τη αλληλεία στην Ευρώπη στο μέλλον. Και αυτή τη στιγμή το κέντρο μοιράζεται με άλλους οργανισμούς όπως το NSA e και τον ε, Παγκόσμιο Θαλάσσιο Οργανισμό δεδομένα. Μια τρίτη πτυχή είναι τα βασικά προγράμματα. Υπάρχουν πρότυπα και ομοιογενές περιεχόμενο σε αυτά τα core curricula, όπως λέγεται, τα βασικά προγράμματα και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί τι συμβαίνει αν αντιληφθούμε παράβαση η οποία έγινε αντιληπτή. και θεώρησα ότι αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να αναφέρω στον εισηγητή για τη μεταρρύθμιση της κοινής ελληνική πολιτικής ότι πραγματικά πρέπει να υποστηρίξουμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον οργανισμό ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα κοινή χρήση των πληροφοριών, ιδίω αυτών που έρχονται από άλλα κέντρα και πιστεύω ότι αυτές οι συμφωνίες ε, ε, συνεργασίας θα μπορούσαν να παρέχουν νομική υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και ο οργανισμός αυτός είναι ένας οργανισμός που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί πλήρως. Θα χρειαστεί κονδύλια λοιπόν για να μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε. Αυτό που είναι πολύ καλό για το κέντρο είναι ότι δεν έχει απλά την αλληλεία. αλλά δοκιμάζει αποτελεσματικά πολίτη σχέδια τα οποία είναι δυνατόν να επαληθευτούν. Αυτά είναι τα όσα μπορούμε να κάνουμε στον τομέα του ελέγχου, του τύπου ε, μελλοντικών προοπτικών που έχουμε σε αυτό το πλαίσιο, στον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κάποιο άλλο να μιλήσει. Όχι, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη. Διακόπτουμε λοιπόν τη συνεδρίαση αυτή μέχρι αύριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη που βρίσκονται ακόμη εδώ που κάτσαν μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 και μετά έχουμε την ε, ημερίδα στις 10.